Liebe Kolleginnen und Kollegen, zuerst einmal einen schönen guten Morgen von meiner Καλημέρα σας. Ε, θα ήθελα να σας ε, πω ότι πριν αρχίσουμε τη συνεδρίαση θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλους να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγής, να σηκωθείτε από τις θέσεις γιατί σήμερα είναι ένας χρόνος από τις επιθέσεις εδώ στις ε, Βρυξέλλες που έγιναν ακριβώς πριν από ένα χρόνο, σχεδόν περίπου αυτή την ώρα. Και να έχουμε λοιπόν ένα, ενός λεπτού σιγή. Herzlichen Dank. Ich möchte Sie ferner... Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι στις 10 μπροστά από την αίθουσα της Ολομέλειας ε, θα υπάρξει μια τελετή από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Βεβαίως ε, είναι δική σα επιλογή να πάτε εκεί. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το σημείο 1 τη ημερήσια διάταξης. Είναι έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Εάν δεν υπάρχουν καθόλου ενστάσει, εγκρίνεται. Σαπίνε. Έχω μία ερώτηση πριν περάσουμε στην ψηφοφορία. Μας είπαν ότι το τμήμα στο ψήφισμα για το Solidarity Corps από την Επιτροπή Απασχόλησης ε, δεν έχει ψηφιστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης. Θα το, πρώτα, θα το διευκρινίσουμε όταν ε, φτάσουμε στη ψηφοφορία εκεί. Θα περάσουμε σημείο 2 της ανακοινώσης της Προέδρου και θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι σήμερα έχουμε μετάφραση στα γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, ισπανικά, τσεχικά, εστονικά, λιθουανικά, πολωνικά, σλοβενικά και ρουμανικά. Ε, και βεβαίως ε, μεταδίδεται από το ίντερνετ η συνεδρίαση. Τώρα η απόφαση των συντονιστών της 27 Φεβρουαρίου σας στάλησαν ε, στις 2 Μαρτίου με email και εγκρίνονται επισήμως εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις δεν υπήρξαν ενστάσεις στις 7 ε, Μαρτίου. Δεν συνέβη, άρα λοιπόν και τα πρακτικά αυτά εγκρίνονται. Και τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Το πρώτο σημείο στην ε, ε, η μέση διάταξη είναι να ψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Σώμα αλληλεγγύη. Αφού ο πρόεδρο Γιούγκερ, όπω ξέρετε, τον προηγούμενο Σεπτέμβριο πρότεινε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ε, και ελήφθησαν κάποια προπαρασκευαστικά μέτρα εκ μέρου Επιτροπής. Οι συντονιστές αποφάσισαν να επεξεργαστούν μια προφορική ερώτηση μαζί με ένα ψήφισμα ε, υποβλήθηκε σε 17 Μαρτίου το προφορικό ερώτημα και συνοδεύεται από μία επιστολή ε, και ε, εγώ επέβαλα την παράκληση να συμπεριληφθεί το ψήφισμα αυτό στην μερίσια διάταξη του Απριλίου και θα ήθελα να παρακαλέσω τους συντονιστές να βρουν να υποστήριξη στις πολιτικές τους ομάδες. Ξέρετε ότι η Κομισιόν το Μάιο θα υποβάλει την νομοθετική της πρόταση για το Ευρωπαϊκό Σώμα Ελεγγύης και στη συνεδρία των συντονιστών όλοι είχαμε την άποψη ότι είναι ε, αναγκαίο και χρήσιμο να υποβάλουμε και τις δικές μας προτάσεις στην ε, Κομισιόν ούτως ώστε να ξεκαθαρίσουμε τι εμείς αναμένουμε από μια τέτοια πρόταση και τι θα έπρεπε να γίνει ε, ενδεχομένω ε, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την χρηματοδότηση ενός τέτοιου Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Η επιστολή πήγε στον πρόεδρο Ταλιάνη δεν μας υποσχέθηκαν τίποτα όσον αφορά την ημερήσια διάταξη γιατί όλα αυτά ε, γίνονται με την επιφύλαξη της απόφασης για το Brexit ε, βάσει του, της του, μετά την ενεργοποίηση του άρθρου 50 κάτι το οποίο βεβαίως θα καθορίσει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Απριλίου. Αλλά πιστεύω ότι ε, έφτασε το μήνυμα ότι για μας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το σημείο. Τώρα θα πράσουμε στην ε, ψηφοφορία για το ψήφισμα. Ε, λόγω της καλής συνεργασίας εντός της Επιτροπής και ε, με άλλες επιτροπές, μεταξύ άλλων της Επιτροπής Απασχόλησης, ε, κάναμε την πρόταση στην Επιτροπή Απασχόληση να μας επισημάνουν από τη δική τους πλευρά ορισμένα σημεία και εμείς ε, ευχαρίστως θα το συμπεριλάβουμε στο ψήφισμά όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Απασχόλησης στον τομέα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Διαβιβάσαμε γέρος αυτή την πρόταση στην Επιτροπή Απασχόλησης και είχαμε και κάποιες προτάσεις χθε το μεσημέρι, αλλά προσπάθησα να τη συμπεριλάβω στο κείμενο στο βαθμό που εμπίπτει στους αρμοδιότητες της Επιτροπής Απασχόλησης και χθε το βράδυ και σήμερα το πρωί μάθαμε ότι προφανώς οι προτάσεις αυτές δεν έχουν ψηφιστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης. Αυτό είναι κάπως δυσάρεστο αλλά να πω και στην διακριτική ευχαίρεια της Επιτροπής Απασχόλησης να αποβάλουν τις προτάσεις τους στην Ολομέλεια. Η πρότασή μου είναι τα σεσημασμένα τμήματα με γκρι ή κίτρινο να τα αφαιρέσουμε απλούστατα. Γιατί όπως σας είπα δεν έχουν ψηφιστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης. Άρα λοιπόν ε, δεν είναι δυνατόν να ψηφιστούν από εμά. Και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η Επιτροπή Απασχόλησης να δει κατά πόσο θέλει να τα προτείνει τα σημεία αυτά στη Ρολομέλη ή όχι. Εγώ θα ήθελα να είχα συμπεριληφθεί, αλλά προφανώς δεν είναι κάτι τέτοιο δυνατόν. Τώρα, όσον αφορά την διαδικασία, Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, κυρίως όσον αφορά στο επίπεδο εργασία. Υπήρξε μια τεχνική συνάντηση και όλες οι τροπολογίες οι οποίες υποβλήθηκαν, γιατί είχαμε συμφωνήσει να υπάρξει μια απλουστευμένη διαδικασία. Να συμπεριληφθούν λοιπόν όλα αυτά στο κείμενο και αυτό το πετύχαμε. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ συνεπές ε, κείμενο και καλό κείμενο και η πρότασή μου είναι να ψηφίσουμε το κείμενο ως έχει στο σύνολό του, εξαιρώντας βεβαίως τα, τις προτάσεις της Επιτροπής Απασχόλησης. Έχετε καμία αντίρρηση να ψηφίσουμε το κείμενο στο σύνολό του. Όχι. Άρα λοιπόν θα περάσουμε στην ονομαστική ψηφοφορία. Ο άλλος κ. Κέστακ μου είπε ότι δεν έχει μαζί την κάρτα του. Θα, θα ε, ψηφίσουμε, θα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Το ψήφισμα αυτό λοιπόν εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ε, συνέβαλαν στην πραγματικά επικοδομητική συνεργασία για, την, ε, για αυτό το ψήφισμα. Και θα δρομολογηθεί η διαδικασία στην Ολομέλεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους δύο αρμόδιους από τις ε, πολιτικές ομάδες και από την, από την γραμματεία, οι οποίοι πραγματικά προσπάθησαν πάρα πολύ για το κείμενο αυτό. Και τώρα θα περάσουμε στην επόμενη ψηφοφορία, που είναι η γνωμοδότησή μας για την έκθεση ε, για την ΕΦΣΥ, την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Συντάκτρια ήταν η Jill Evans και οι συνάδελφοι ε, πρότειναν να γίνει συμφωνία μέχρι τον Ιούνιο. Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα ε, νωρίτερα από ό,τι είχε αποφασιστεί το σχέδιο υποβλήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου, οι τροπολογίες στις 3 Μαρτίου, υπάρχουν 22 τροπολογίες και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες για την αποκαδομητική ε, συνεισφορά τους. Και θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Evans εάν θέλει να πάρει το λόγο πριν από την ψηφοφορία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας ευχαριστήσω καταρχάς ε, για τα, για τα σχόλιά σας για το χρονοδιάγραμμα. Τα πράγματα ήταν βέβαια έτσι πιο δύσκολα, αλλά ήταν πολύ καλή συνεργασία μας. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους κοιότητες εισηγητές, τα μέλη της γραμματείας, ε, το δικό μου ε, προσωπικό και το προσωπικό της ομάδας μου, γιατί καταφέραμε νομίζω να συνεργαστούμε καλά και να καταλήξουμε σε μια πολύ καλή γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα περάσουμε στη ψηφοφορία. Θα ξεκινήσουμε την τροπολογία παριθμών 1. Υπέρ παρακαλώ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2. Υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3. Υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμό 1. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα έρθουμε στην τροπολογία παριθμών 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία υπαρθμών 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές νομίζω θα πρέπει να γίνει επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία Πέρας της ψηφοφορίας. 12 προς 12 απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά αν θέλετε να γίνει έλεγχος λοιπόν μόνο 19 τροπολογία άρχεται η ψηφοφορία Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα θα περάσουμε στην τελική ψηφοφορία, είναι ονομαστική, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας, με μεγάλη πλειοψηφία, 22 ναι, ένα όχι, μία αποχή, θερμά συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Και τώρα το σημείο 5 της ημερήσία διάταξης. Εδώ πρόκειται για μια γνωμοδότηση της Επιτροπής μας για το φόρο προστιθέμενες αξίας για βιβλία, εφημερίδες, ε, περιοδικά κλπ. Η συγητής είναι ο συνάδελφος Τρογεύσκη Του δίνω το λόγο. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για μια γνωμοδότηση πολύ σημαντική. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα επίσης. Αφορά το ΦΠΑ, το ποσοστό του ΦΠΑ και πρόκειται για μία μάχη πάνω από 10 ετών σε σχέση με την ηλεκτρονική δημοσίευση, ε, τα ηλεκτρονικά ε, βιβλία δηλαδή να ε, εισάγονται με μειωμένο ποσοστό ΦΠΑ. Ξεκίνησε από ένα ευρύτερο πακέτο. Πρόκειται για μία εναρμόνιση των διατάξεων σε θέματα ΦΠΑ στην ψηφιακή οικονομία. Έχουμε δύο χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, που δεν συμφωνούν με υψηλότερα ποσοστά ΦΠΑ ε, όσον αφορά την ψηφιακή οικονομία και την ηλεκτρονική δημοσίευση. Υπάρχουν μάλιστα προσφυγές που έχουν γίνει ενώπιον των δικαστηρίων και εμείς εδώ απαντούμε στις ε, διάφορες προσδοκίες όσων θα ήθελαν όλα αυτά να είναι εναρμονισμένα και να υπάρχουν προτιμησιακά ποσοστά στις ε, δημοσιεύσεις ε, βιβλίων ηλεκτρονικά. Έχουν ήδη μειωμένο ποσοστό ΦΠΑ και στις δύο περιπτώσεις λοιπόν υπάρχουν διαφορές Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μεταχειριζόμαστε ε, ε, ε, ένα προϊόν ως προϊόν και άλλες περιπτώσεις όπου το μεταχειριζόμαστε ως υπηρεσία. Τα κράτη-μέλη πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν το ίδιο ποσοστό μειωμένου ΦΠΑ και για τα περιοδικά και για τα βιβλία τα ηλεκτρονικά και το ίδιο ισχύει και, για τις, και, με, τις, με τις δημοσιεύσεις τις έντυπες. Αυτές οι δημοσιεύσεις είναι υπηρεσίες που ε, παρέχονται μέσω ε, ηλεκτρονικής οδού και έχουν ε, ένα ποσοστό φόρου διαφορετικό. Εμείς δεν έχουμε αμφιβολία ότι θα έπρεπε να γίνει εναρμόνιση αυτών των ποσοστών και να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να μειώσουν το ποσοστό ΦΠΑ τους. Πρόκειται λοιπόν για μια πρόταση η οποία είναι καλή είναι πολύ θετική η άποψή μας, είναι πολύ λίγες οι προτάσεις τροπολογιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ε, συντάξτες αυτών των τροπολογιών και δέχομαι με πολύ χαρά όλες αυτές τις προτάσεις που γίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να κλείσουμε και αυτές τις ε, ε, προσφυγές και αυτή την τόσο μακρόχρονη σύγκρουση. Ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι αυτή είναι μια σχεδόν ατέρμονη ιστορία, αλλά τελικά όλα βαίνουν καλώς. Και κανείς ε, δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί θα πρέπει για μια έντυπη εφημερίδα να πληρώσει λιγότερο ΦΠΑ από ότι ε, για μια εφημερίδα στο ίντερνετ. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι ότι όλα αυτά τώρα διατυπώνονται γραπτά και ελπίζω ότι αυτή η ιστορία θα ε, έχει θετική έκβαση και θα υποβάλλει αντιστοίχω και η Κομισιόν τη δική της πρόταση. Τώρα, η Σκιώδης, ο κύριος Μοργάνο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον ε, εισηγητή Σδρογεύσκη για την εξαιρετική έκθεση και για αυτή την προσέγγιση η οποία στην ουσία ε, οδηγεί σε μια εξισορροπημένη τελική πρόταση. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολούσε εδώ και καιρό στο Κοινοβούλιο, ήδη από το 2011. Ξέρουμε ότι το βιβλίο είναι βιβλίο, το περιοδικό περιοδικό. Ε, είναι μια φυσική οντότητα, όχι όπως ε, το διαδίκτυο και η ταμπλέτα. Παρόλα αυτά, στην ψηφιακή εποχή θα πρέπει να άρουμε αυτή την διάκριση που είναι απαρχαιωμένη και να μιλάμε για προϊόντα που έχουν ιδιαιτερότητες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τους νέους, οι οποίοι χρησιμοποιούν ε, το ψηφιακό περιεχόμενο και για δημιουργικούς σκοπούς και για σκοπούς αναψυχής ή εκπαίδευσης για τη διάδοση του πολιτισμού με λίγα λόγια. Άρα έχουμε θετικές συνέπειες από ότι προβλέπεται από αυτό το πλαίσιο και αυτό σε σχέση με την φορολόγηση η οποία θα πρέπει να ε, μειωθεί και να φτάσει στη μηδενική. Οι εκδότες λοιπόν δεν θα πρέπει να εξαρτώνται τόσο πολύ από τη διαφήμιση. Σημερίζομαι την προσέγγιση του εισηγητή και ε, έχω υποβάλει μόνο δύο τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη. Και εγώ θα υποβάλω δύο τροπολογίες ε, συμπληρωματικού χαρακτήρα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εγκριθεί τάχιστα αυτή η έκθεση και προσέγγιση από το Συμβούλιο Υπουργών. και από πλευρά τη άλλη επιτροπή θα συνεισφέρω επίσης. Uh, Ευχαριστώ. Μιλώ σήμερα εκ μέρου ε, του Τζον Fox και νέου συναδέλφου, ο οποίο δυστυχώ δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο γιατί έχω πολλέ ε, τέτοιου είδου αντικαταστάσει να κάνω σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή για την ε, καλή του γνωμοδότηση και επειδή ε, δέχτηκε αυτέ τι δύο τροπολογίε για την καινοτομία που εμεί ω ECR ευχαρίστω θα υποστηρίξουμε. Επίση έχουμε την τάση να συμφωνούμε με την γενική κατεύθυνση τη Επιτροπή που λέει ότι πρέπει να υπάρχει ευελιξία σε εγχώριο ΦΠΑ ανάλογα με τι συνθήκε και τις ανάγκε και στις περιπτώ... η μόνη περίπτωση στην οποία θα είχαμε κάποιου ενδιασμού είναι όταν αυτό μπορεί να ε, διαστρεβλώσει τον ε, ανταγωνισμό. Πάντω σε γενικές γραμμέ, συμφωνούμε με τι απόψει που ε, εκφράζει αυτή η γνωμοδότηση. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και οι πράσινοι υποστηρίζουν αυτή την πρόταση και θεωρώ θετικό ότι πηγαίνουν τα πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση. Το κόστος για τα βιβλία και το ίντερνετ ε, μειώνεται. Είναι σημαντικό ε, και το Κοινοβούλιο να συνεργαστεί εδώ. Στην ε, Αυστρία δεν υπάρχει ομοφωνία ε, για το θέμα αυτό. Εάν ε, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συνεργαστούν, έχουμε μια πιθανότητα να περάσει και αυτό στις άλλες ε, χώρες. Νομίζω θα ήταν καλό βεβαίως να επισημάνουμε ότι κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανόνες, αλλά εάν μπορούμε να μειώσουμε ενιαία το κόστος ε, αυτό θα είναι ένα πολύ θετικό βήμα, αλλά βεβαίως ε, θα πρέπει να πιστεί και το Συμβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Πέλτ. Euh, Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Η, η πρόταση του Συμβουλίου νομίζω ότι πηγαίνει προ σωστή κατεύθυνση γιατί δίνει μεγαλύτερη ελευθερία στα κράτη-μέλη για την επιβολή ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, ε, το μειωμένο ποσοστό ε, το 5,5% δίνει τη δυνατότητα μιας, ε, ε, την οικονομία, της οικονομίας ηλεκτρονικής των βιβλίων να ανθίσει. 91% των Γάλλων διαβάζουν τα βιβλία αυτά και χαίρομαι ιδιαίτερα που το μειωμένο αυτό ποσοστό θα ισχύσει και για τα ηλεκτρονικά βιβλία γιατί το, από το 2012 το κάνει αυτό η Γαλλία και έχει μάλιστα συγκρουστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήθελε να ε, μην ε, Ισχύει αυτό το μειωμένο ποσοστό. Ένα ε, βιβλίο αποτελεί ένα βιβλίο, όποιο και αν είναι το μέσο που χρησιμοποιούμε. 22% των Γάλλων χρησιμοποιούν τα βιβλία αυτά τα ηλεκτρονικά. Θα ήθελα να αναφερθώ στην γνωμοδότηση του συναδέλφου, να τον ευχαριστήσω κιόλας, γιατί μέσω των τροπολογιών του είπε πόσο σημαντικό είναι ε, να υπάρχουν απαιτήσει ε, προσβασιμότητας ε, για άτομα με αναπηρίες. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ο hm? κύριος Χουντής, συγγνώμη. Κυρία Πρόεδρε, ε, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας ε, για την προσπάθεια που κατέβαλε. Φαίνεται ότι λύνεται ένα πρόβλημα που μας απασχολούσε, απασχολούσε όλα τα κράτη, αλλά και κάθε Ευρωπαίο πολίτη με ευαισθησίες στα πολιτιστικά, στην ε, πρόσληψη πολιτιστικών ε, προϊόντων. Ε, φαίνεται ότι λύνεται, επαναλαμβάνω. Γενικώ έχουμε το φαινόμενο γενικώς του προβλήματος του ΦΠΑ ή και εν γέννη της φορολογίας που σε περίοδο κρίσης πολλές φορές λειτουργεί αποτρεπτικά για να προσέλθει ο εργαζόμενος, ο πολίτης που έχει περιορισμένα οικονομικά σε αυτά, δηλαδή μειώνονται οι πωλήσει τουλάχιστον των παραδοσιακών βιβλίων σε γενικές γραμμές και επομένως αυτή είναι μια πρώτη προτεραιότητα και οι δικές μου παρατηρήσεις λοιπόν είναι ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των πολιτών ε, και πολιτών που έχουν ε, σε οικονομικά προσβάσιμα βιβλία και έντυπα και ηλεκτρονικά και αυτό πρέπει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Νομίζω το, τονίζει ο εισηγητής, συμφωνώ λοιπόν με αυτό. Και η δεύτερη, ε, ας το πούμε έτσι, παρατήρηση που έχω να πω είναι ότι το γεγονός ότι εξισώνονται οι συντελεστές ΦΠΑ ανάμεσα στις κλασικές και στις ηλεκτρονικές εκδόσεις μπορεί να δημιουργήσει βραχυπρόθεσμα τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες για την ανάπτυξη του κλάδου, αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως, και δεν μπορεί βεβαίως ο εισηγητής να το λύσει αυτό το πρόβλημα, ότι θα έχουμε μείωση των τελικών τιμών, μείωση των τελικών ε, τιμών και ε, αύξηση της πρόσβασης των πολιτών ε, μακροπρόθεσμα. Το επαναλαμβάνω για να γίνω κατανοητός. Βραχυπρόθεσμα θα δώσει μια όθωση στον κλάδο, αλλά μακροπρόθεσμα δεν μπορεί να το προβλέψει, ούτε μπορεί να το ελέξει ότι θα το έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που είναι σωστό στόχο και σωστή επιθυμία. Επομένω, το ζητούμενο είναι να μπορέσουν να διασφαλιστούν η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, ούτω ώστε να αντικατοπτρίζεται άμεσα η μείωση των συντελεστών να αντικατοπτρίζεται και στις τιμές των ηλεκτρονικών εκδόσεων και να μην αποτελεί μια ιδιαίτερη ευνοϊκή μεταχείριση στους α, ε, ε, παραγωγούς τέτοιων εκδόσεων. Ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη ομοφωνία εδώ στην αίθουσα. Θα ήθελα παρόλα αυτά να ρωτήσω την Επιτροπή αν θέλει να πάρει το λόγο. Κύριε Φαντίνη, παρακαλώ. Bitte, Sie haben um, Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για την έκθεση αυτή που ε, στην ουσία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας και τη διασύνδεσή της με την ε, ψηφιακή πρωτοβουλία Η πρωτοβουλία αυτή συζητείται στο Συμβούλιο επί της παρούσης και ελπίζουμε να εγκριθεί σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και θα ήθελα να σας επισημάνω ότι η βάση για αυτή την... η νομική βάση είναι το άρθρο 130. Θα υπάρξει διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, αλλά ελπίζουμε ότι μέσω της ε, διαβούλευσης θα αποστείλουμε ένα γρήγορο μήνυμα προς το Συμβούλιο, ούτως ώστε να πετευθεί τάχιστα η συμφωνία. Προθεσμία 28 Μαρτίου στις 11 για την υποβολή τροπολογιών οι τροπολογίες κατ' εξαίρεση μπορούν να υποβληθούν μόνο στα αγγλικά. Αυτό έχει να κάνει με τις ημερομηνίε. Αλλά νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή δεν είναι τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό και θα πρέπει να υποβληθούν μέσω της γραμματείας, όχι όπως ε, βάσει του συνήθου συστήματος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση αυτή και θα περάσουμε άμεσα στο επόμενο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρα της βιωσιμότητας. Η συγκέντρια είναι η συνάδελφος ε, Λιάντ Νιριάντα η οποία δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα στη συνεδρίαση και γι' αυτό ο κύριος Χουντής θα παρουσιάσει εκ μέρους της την έκθεση. Παρακαλώ κύριε Χουντή. Ε, σας ευχαριστώ και πάλι κυρία Πρόεδρε. Ε, όπως είπατε αγαπητοί συνάδελφοι, η συνάδελφος εισηγήτρια της σχετικής γνωμοδότησης ε, απουσιάζει, είναι στην κηδεία του Μαγκίνες στην Ιρλανδία. Με παρακάλεσε να παρουσιάσω εγώ εκ μέρους της τη γνωμοδότηση ε, θα το αποπειραθώ, θα είμαι σύντομος, αλλά θα σεβαστώ και το γραπτό κείμενο για να μπορέσω να αποδώσω σωστά τις σκέψεις της, ε, ε της εισηγήτριας. Την γνωμοδότηση την έχετε δει. Το θέμα το θεωρεί η εισηγήτρια και εγώ βεβαίως και εμείς εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ίσως είναι και βασική πλευρά της δράσης της Επιτροπής μας. Από τις βασικότερες πλευρές της δράσης της Επιτροπής μας. Ε, θα ήθελε να περιλάβει αρκετά στοιχεία κατά συνέπεια, αλλά λόγω του περιορισμένου χρόνου, εντός των ορίων πρέπει να κινούμεθα στις γνωμοδοτήσεις, επέλεξε να βάλει, <clears throat> συγγνώμη, επέλεξε να τονίσει πέντε βασικούς τομείς, όπως φαίνονται και από τις σχετικές παραγράφους του κειμένου που έχετε μπροστά σας, της σχετικής γνωμοδότησης. Το πρώτο είναι ότι πιστεύουμε ότι για την προετοιμασία ενός βιώσιμου μέλλοντος και για την αντιμετώπιση των οικονομικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων η ύπαρξη ποιοτική και χωρί αποκλεισμού εκπαίδευση και διαβίου μάθηση για όλου αποτελεί προαπαιτούμενη συνθήκη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό χαιρετίζει την υιοθέτηση του θεματολογίου 2030 για την αεφόρο ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα το στόχο 4 από την 70η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού ΟΗΕ. Επίσης σημειώνει ότι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καυχάται του πρωταγωνιστή σε αυτούς τους θα πρέπει να είναι να ενσωματώσει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης της πολιτικές της. Στο σημείο 2 τονίζεται ότι για να επιτευχθεί ο στόχος 4 ε, είναι απαραίτητη η επαρκή χρηματοδότηση των δημοσίων συστημάτων εκπαίδευσης. Σε αυτό το σημείο, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Επιτροπής, η εισηγήτρια εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι μεταξύ 2010 και 2014 οι επενδύσεις στην εκπαίδευση έπεσαν κατά 2,5 στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Είναι σημαντικό να γίνει σαφές ότι η υιοθέτηση τέτοιων φιλόδοξων στόχων πρέπει να εξασφαλίσουν και την απαραίτητη δαπάνη. Ένας αστερίσκος από τη δική μου την πλευρά, οι χώρες που βρίσκονται σε μνημόνιο όπως η χώρα μου, αλλά και μια τάση γενικής λιτότητας περικοπής κοινωνικών δαπανών, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό που επισημαίνεται εδώ και που νομίζω ότι μας απασχολεί όλους η μείωση των δαπανών. Το τρίτο σημείο είναι <clears throat> ότι για να μπορέσουν να επιτευχθούν ε, χωρίς αποκλεισμούς ισότιμη ποιότητα της εκπαίδευσης και πρόθεση των ευκαιριών διαβίου μάθησης <clears throat> για όλους, χρειάζεται μια συνολική αναθεώρηση των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ε, αυτό τονίζει η συγήτρια στο τρίτο σημείο. Ε, αυτή η αναθεώρηση θα πρέπει να βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και θα αποσυνδέει από την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των συμφερόντων της αγοράς. Στο κείμενο τονίζεται και νομίζω εδώ δεν πρέπει να έχουμε ε, διαφωνία ότι το θέμα της ε, εκπαίδευσης και το θέμα των δεξιοτήτων δεν είναι ένα θέμα που πρέπει μονόπλευρα να συνδέεται μόνο με το θέμα της ε, αγοράς εργασίας αλλά ότι αυτές οι διαδικασίες πρέπει να προωθούν κατά ολιστικό τρόπο, δηλαδή κατά καθολικό τρόπο ή κατά πολυδιάστατο τρόπο την, οικονομική, την προσωπική συγγνώμη, και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου επομένως έχει μια αυταξία. Αυτό τονίζει το σημείο 3. Το σημείο 4 και το πρώτο τελευταίο, ότι πρέπει να υπάρξει βέλτιστη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων. Αυτό μας έχει απασχολήσει ε, από την παρακολούθηση και τη συμμετοχή στην Επιτροπή, το έχω δει και σε άλλες περιπτώσεις, και να υπάρχουν συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων, όπως παραδείγματο χάρη το Erasmus+, Plus, και σε μια τέτοια περίπτωση αυτές οι συνέργειες πρέπει να αποδώσουν βελτίωση και εξυγχρονισμό στην ποιότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και επίσης τονίζει την ανάγκη να αρθεί κάθε αποκλεισμό από τους κατοίκους των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών από τις δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης, μια κατάσταση η οποία επικρατεί λίγο πολύ σε όλες τις χώρες σε σχέση με τις δυνατότητες των κατοίκων σε αυτές τις περιοχές. Και τέλος, η εισηγήτρια αναφέρεται στο διαρκές πρόβλημα της ανεργίας των νέων, που σε ορισμένα κράτη-μέλη αγγίζει το 40%, βάζω την πινελιά την ελληνική, στην Ελλάδα ξεπερνάει το 50% πρωταθλήτρια στην ανεργία των νέων, αλλά και σε αρκετέ χώρε του Νότου αυτό το ποσοστό είναι παραπάνω από το μέσο όρο που εμφανίζεται γενικώ στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα αυτά, ε, το πρόγραμμα τονίζεται στην γνωμοδότηση ότι το πρόγραμμα, τα προγράμματα για τις εγγυήσεις για την νεολαία και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων αδυνατόν να δώσουν βιώσιμες λύσεις για τους νέους και προτείνει την αναθεώρησή τους με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας και την πρέπουσα κοινωνική προστασία των νέων. Ε, αυτά είχα να πω εκ μέρους της εισηγήτριάς μας. Είπα και εγώ ορισμένες πινελίες. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ja, vielen herzlichen Dank. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα πάρουν το λόγο οι εγώ γνωρίζω μόνο τους δύο ονομαστικά. Δεν ξέρω εάν κάποιος ε, άλλος επιθυμεί από κάποια άλλη πολιτική ομάδα. Παρακαλείτε να πάρει το λόγο, η Τζούλι Γουότ. Μπορώ να ε, μιλήσω αργότερα, Πέτρα, γιατί ξέχασα τις σημειώσεις μου και η Τζούλη έτρεξε να μου τις φέρει. Μπορεί να λάβει το λόγο κάποιος άλλος. Τότε Τότε, κυρία Μπιλ. Ευχαριστώ. Αναμφισβήτητα υπάρχουν θετικά στοιχεία σε αυτή την ε, γνωμοδότηση της κυρίας Ριάντα. Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει η ίση η πρόσβαση στην εκπαίδευση στις απομακρυσμένες περιοχές, στις αγροτικές περιοχές. Δυστυχώς 11.000 τάξεις έκλεισαν στην ε, Γαλλία. Αυτή η απερίμωση του αγροτικού ε, κόσμου οδηγεί σε μία έξοδο, μαζική έξοδο προς τα αστικά κέντρα. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μία ε, επίλυση του ζητήματος με τα γειτονικά σχολεία. Αυτό έχει σχέση και με την απασχόληση των νέων. Δυστυχώς οι λύσεις θα πρέπει να κινούνται προς τα πάνω. Αυτό αφορά και την κατάρτιση και την επαγγελματική εκπαίδευση που γίνεται πολύ αργά. Επειδή υπάρχουν θέματα βιωσιμότητας, θα ήθελα να γίνει λόγος για την πολιτική αγωγή τη διδασκαλία της πολιτικής αγωγής στα σχολεία. Θα υποβάλω τροπολογίες επί του θέματος. Ευχαριστούμε. Η Julie Watts έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα για μένα. Ήμουν φοιτήτρια και στη συνέχεια ασχολήθηκα ε, με αναπτυξιακά θέματα, ιδιαίτερα στο SDG ε, Watch. Εκεί εργάστηκα για να δω ε, κατά πόσο μπορούμε να φτάσουμε και στους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Μιλήσαμε λοιπόν για τη βιωσιμότητα και την εκπαίδευση κυρίως και στο, στην πτυχιακή μου ιδιαίτερα ασχολήθηκα με αυτό το θέμα. Υπάρχουν τρεις ε, πυλώνες, ε, ο οικονομικός, κοινωνικός και ο περιβαλλοντικός. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να φτάσουμε σε μία στοχοθέτηση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει συστηματικός τρόπος για να φτάσουμε σε ένα πολιτισμικό αναπτυξιακό πρότυπο. Δυστυχώς, λοιπόν, στην έκθεση αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος κλειδί του πολιτισμού. Νομίζω, λοιπόν, ότι η έκθεση είναι ελλειπής σε αυτό το στάδιο. Υπάρχει και ο πολιτισμικός πυλώνας για μένα, ε, ο οποίος είναι φορέας δημιουργίας νέων τρόπων ζωής και παραδειγματικών τρόπων ζωής. Αυτό σημαίνει να υπάρχει μια τοπική κατανόηση της ε, συλλογικής ανάπτυξης. Εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ρόλο του πολιτισμού ως ε, διευκολυντή ώστε να φτάσουμε και στους περιβαλλοντικούς στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Άρα, ο πολιτισμός είναι φορέας ανάπτυξης και καινοτομίας μέσα στα πλαίσια των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και συλλογικής ευημερίας. Είναι ύψης της σημασίας για να λάβουμε υπόψη την ολιστική προσέγγιση του ζήτηματος και να μην κινηθούμε με στεγανά. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να ληφθούν υπόψη από τους πολιτικούς. Γι' αυτό θα πρέπει το Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με, το, με τους SDG, δηλαδή τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης συνολικά και οριζόντια. Όταν μιλάμε για αυτή την ε, ολιστική προσέγγιση, θα ήθελα να μιλήσουμε και για τη συμμετοχή των δύο φύλων, gender mainstreaming, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, την κοινωνία των πολιτών, την έρευνα και συλλογή στοιχείων, αποδεικτικών στοιχείων έτσι ώστε να μιλήσουμε για τη σχέση μεταξύ επιστήμων και πολιτισμού. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μία συλλογική σκέψη και συλλογιστική επί του θέματος. Αυτό το βλέπουμε και στις τέχνες ιδιαίτερα που θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη στο, στο δημόσιο χώρο μας. Έτσι μπορεί η ζωή να γίνει πιο βιώσιμη χωρίς αποκλεισμούς. Έτσι ώστε να βάλουμε τον άνθρωπο στον, στο επίκεντρο του γενικότερου μελήματός μας. Ευχαριστώ πολύ, Helga Trüppel. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τα βασικά θέματα που έθεξαν η Τζούλη και ο συνάδελφος κ. Χουντής. Νομίζω ότι οι λεπτομέρειες ε, δεν είναι καινούριε. Έχουμε συζητήσει το θέμα των ε, διεξιοτήτων, εράσμους Plus ε, και λοιπά και τους στόχους της ανάπτυξη. Αλλά βεβαίως το θέμα είναι όλα αυτά να συμπεριληφθούν σε μια κοινή στρατηγική. Αλλιώς δεν θα είναι παρά μια επανάληψη θεμάτων τα οποία έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ε, δεν είναι κάτι καινούριο στο επίπεδο του περιεχομένου. Αλλά θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι θέλουμε να, είναι μια, να υπάρξει μια στρατηγική προσέγγιση. Ε, και πάλι ε, δεν θα έπρεπε να υπάρξουν επαναλήψεις θεμάτων που έχουν ήδη συζητηθεί. Η στρατηγική πτυχή θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ευχαριστώ πολύ η Κομισιόν. Εκτός αν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Ευχαριστώ πολύ, Πέτρα. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρατήρηση και στην Επιτροπή Ανάπτυξης προσπαθούμε να επεξεργαστούμε μια, ένα νέο μοντέλο για την ε, ανάπτυξη. Και ίσως εδώ κατά ε, ε, και, η Προεδρία της Μάλτας ε, συμφωνεί να συμπεριληφθεί ο πολιτισμός εδώ. Βεβαίω θα πρέπει κάποια πράγματα να διευκρινιστούν. Συμφωνώ με τη Τζούλη και εάν θέλουμε να συμπεριλάβουμε τους στόχους, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ε, δεν θα πρέπει να παραμελήσουμε την, ε, τον πολιτισμό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντέβα, εκ μέρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κύριε Βαντρουγκίν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ε, άκουσα συγκεκριμένες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα όμως ε, να μιλήσω για το ανακοινωθέν της Επιτροπής της 21 ε, Νοεμβρίου πέρσι, όπου μιλήσαμε για την εφαρμογή των SDGs, των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και θα ήθελα να σας πω ότι το ανακοινωθέν και ανακοινωθέν αυτό μιλά για την καλύτερη ρύθμιση του ζητήματος έτσι ώστε να ε, εξασφαλίσουμε τους, βιώσιμους, ε, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης από όλες τις ε, πλευρές να έχουμε τη βέλτιστη δυνατή προσέγγιση του ζητήματος και γενικότερα μία ολιστική προσέγγιση έτσι ώστε να καταρρύψουμε τα στεγανά που υπάρχουν. Και βεβαίως να ε, λάβουμε υπόψη την εκπαίδευση και τον πολιτισμό και το συσχετισμό τους. Αν υπάρχουν ε, πιο ειδικέ ερωτήσεις θα είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω άμεσα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να παρακαλέσω την εισηγήτρια, την εκπρόσωπό ε, ή τον εκπρόσωπό της να πάρει πάλι το λόγο. Κύριε Χουντή, παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Παρά το γεγονός ότι δεν είμαι ο εισηγητής, ε, αντιλαμβανόμενος το θέμα κατά τον τρόπο που το αντιλαμβάνεται η εισηγήτρια βεβαίως, η συζήτηση που, και οι παρατηρήσεις που ακούστηκαν από τους συναδέλφους Σκιώδη και άλλου εισηγητέ έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και επομένως αυτό που μπορώ να πω εγώ, συνοψίζοντας ίσως τη συζήτηση ή μια παρατήρηση, οι παρατηρήσει που έγιναν οι επιμέρους και οι τροπολογίες θα κατατεθούν, θα τι δει η ίδια η εισηγήτρια πώς θα τις επεξεργαστεί. Ε, θέλω να σας πω μόνο ότι ε, οι παρατηρήσει που έγιναν για ενδεχόμενες ελλείψεις του κειμένου ή για τη μη συμπερίληψη με μεγαλύτερη σαφήνεια του πολιτισμού μέσα σε όλο το πλαίσιο της, ε, της γνωμοδότησης ε, απαντείται, από μια πλευρά από την εισαγωγική παρατήρηση ότι ο περιορισμένος χρόνος δεν δίνει τη δυνατότητα να αναφερθεί σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει αυτό το θέμα, δηλαδή η ικανοποίηση των στόχων για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το ένα είναι αυτό. Ε, δεν αποτελεί δικαιολογία, αλλά θέλω να πω πώς το καταλαβαίνω, διότι είναι πράγματι σοβαρή παρτής. Και η δεύτερη είναι μια γενικότερη συζήτηση. Θέλω να πω ότι οι προτεραιότητες που έθεσε η συγγήτρια και παρουσίασα εγώ στο κείμενο ε, έχουν σχέση με τη συγκεκριμένο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής και σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, η επισήμαση ορισμένων προβλημάτων που έχουν ε, χαρακτήρα, με το θέμα της εκπαίδευσης, με το θέμα των νέων, υπαγορεύεται από αυτή την συγκυρία της προτεραιότητας. Κατά τα άλλα, η συζήτηση για τον αναπτυξιακό ρόλο του πολιτισμού έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό είπα ότι ε, ε, θα ήθελα να περιλαμβάνετε, αλλά προσπαθώ να σας πω γιατί όπως κατάλαβα και εγώ, η εισηγήτρια επέλεξε αυτά τα θέματα να σταθεί. Δεν σημαίνει ότι αγνοούσε τη σημασία ή δεν σημαίνει ότι η παρατήρηση των συναδέλφων, της συναδέλφων, των συναδέλφων δεν έχουν καμιά αξία και επομένως ε, θα απορριφθούν κτλ. Ε, εγώ αυτά ήθελα να πω. Θα μεταφέρω τις παρατηρήσεις και ε, τη συζήτηση στην εισηγήτρια η οποία θα τελειώσει το έργο της με τη δική μας στήριξη όλων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 29η Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι και η ψηφοφορία θα γίνει στις 25 Απριλίου στην Επιτροπή Πολιτισμού. Ευχαριστούμε πολύ. Με μεγάλη χαρά θα ήθελα να καλωσορίσω μία ομάδα επισκεπτών που προσεκάλεσε ο κ. Μαλινόφ από το Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο στο Παρίσι. So, wir. από το Βουλγαρικό Σχολείο, συγγνώμη, στο Παρίσι. Και τώρα θα έρθουμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης θεμητά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον όταν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών. Η συγκητής είναι ο κύριος Κρασνοντέψκι και θα γνωρίζετε ότι εδώ και 1,5 χρόνο στο Κοινοβούλιο γίνονται έντονες συζητήσεις εν σχέση με τις ενότητες αποτελεσματικής προστασίας των ε, καταγγελτών. Για παράδειγμα, δημοσιογράφους, ε, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την προστασία των πηγών εδώ. Και υπάρχει μια πρόταση Ο κύριος Λούα θα εκπροσωπήσει τον κύριο Καζνοτεύσκη και του δίνω μέσο στο λόγο. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε. Ναι, εκπροσωπώ τον κύριο Καζνοτεύσκη και θα ήθελα να σας αναφέρω τις σκέψεις τους από την ε, οπτική γωνία της Επιτροπής μας. Η σημασία της προστασία των καταγγελτών έγινε προφανής ε, τα τελευταία χρόνια όπου υπήρξαν πάρα πολλές ε, παράτυπες αποκαλύψεις Panama Leaks, Swiss Leaks κλπ. Ε, και ε, με τις εργασίες Επιτροπής Τάξ έγινε προφανές ότι είναι σημαντικός ο ρόλος των καταγγελτών όσον αφορά την αποκάλυψη δραστηριοτήτων που παραβιάζουν το δημόσιο συμφέρον. Ε, ωστόσο, οι καταγγελίες είναι όσον αφορά τις οικονομικές αποκαλύψεις, είναι ο μόνος μηχανισμός αποκαλύψεων. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός προστασίας για καταγγέλλοντες οι οποίοι ε, καταγγέλνουν τις λειτουργίες στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ε, πρόθεση είμαστε να εστιάσουμε σε τρεις ε, στόχους που εμπίπτουν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Στα, τα θέματα αυτά αφορούν καταρχήν πολιτιστικές διαφορές στην πρόσληψη των καταγγελτών. Επίσης, ε, πρωτοβουλίες εκπαίδευσης ε, που να ενθαρρύνουν τις διαδικασίες αυτές ε, καταγγελίες. Επίσης, είναι σημαντικό να, οι μηχανισμοί προστασίας των καταγγελιτών να είναι προσαρμοσμένες στις καταστάσεις που επικρατούν στις διάφορες χώρες μέλη, στις πολιτιστικές διατεστερότητες της κάθε χώρας. Γιατί οι εσωτερικές διαδικασίες ε, εντός των θεσμικών οργάνων ε, καμιά φορά συνδέονται με προβλήματα και τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το ίδιο ισχύει όσον αφορά εθνικά μέτρα προστασίας συστημάτων καταγγελίας. Βεβαίως, η αναφορά σε πολιστικές ε, ιδιαιτερότητες δεν θα πρέπει να χρησιμεύσει ως άλοθη για την έλλειψη προστασίας. Απλώς οι ίδιοι μηχανισμοί θα πρέπει να αντανακλούν τις πολιστικές διαμορφωγίες. Ε, για παράδειγμα, σε ένα πολιστικό πλαίσιο, ε, η ιδέα μιας οικονομικής επιβράβευσης του εκαταγγέλλοντος μπορεί να βρει απήχηση. Ενώ σε άλλες χώρες υπάρχει τεράστια αντίσταση όσον αφορά αυτό το σύστημα επιβράβευσης. Υπάρχουν χώρες όπου υπάρχει μια γενικά αρνητική πρόσληψη των καταγγελόντων και του μηχανισμού καταγγελίας. Άρα το κοινωνικό περιβάλλον είναι μη ευνοϊκό. Άρα θα πρέπει να υπάρξει θέσπιση νομικών διαδικασιών, η οποία όμως να συνοδεύεται από εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που προάγουν την διαδικασία καταγγελίας ως στο κομμάτι μιας ε, σωστής τάσης εκ μέρους των πολιτών. Ε, θα πρέπει να δοθεί έμφαση ότι εσωτερικέ διαδικασίε καταγγελίες δεν θα πρέπει να εξυπηρετούν τον περιορισμό της ελευθερίας του λόγου ή τον περιορισμό της πρόσβασης του κοινού σε σημαντικές πληροφορίες. Σημαντική είναι η διασύνδεση επίσης με, με την ερευνητική δημοσιογραφία. Ο ρόλος των δημοσιογράφων εξαρτάται βεβαίως από την ε, πρόθεση των εργοδοτών να αποκαλύψουν κάποιες ε, ατασταλίες. Ε, και είναι σημαντικό για τις χώρες μέλη να, να εξασφαλίζουν ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν να ασκήσουν ελεύθερα τη δουλειά τους χωρίς να αποκαλύπτουν τις ε, πηγές πληροφόρησης. Για να καταλήξω θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι προκειμένου να υπάρξει μια προσθέμενη αξία θα πρέπει να αποφύγουμε τις ε, συγκρούσεις συμφερόντων ε, με τις άλλες επιτροπές και θα ήθελα να επαναλάβω ότι υπάρχουν πολιτικές διαφορές όσον αφορά το ρόλο των καταγγελτών θα πρέπει να υπάρχει ελευθερία λόγου για τους δημοσιογράφους όσον αφορά την έρευνά τους. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα τώρα να δώσω το ρόλο στους σκιώδεις για δύο ή τρία λεπτά γιατί δεν έχουμε πλέον τόσο πολύ χρόνο και θα ήθελα να ξεκινήσω εκ μέρους του ΕΛΚ με την κυρία Ζαντρόβα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο Κρασνοντέμσκι για το σχέδιο γνωμοδότησή της. Εγώ μπορώ να συμφωνήσω καταρχήν. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό ε, το γενικό πλαίσιο. Φυσικά υπάρχουν ε, διαφορές ε, απόψεων Πρόκειται για ένα από τα βασικά μέσα που υποστηρίζει την πρόληψη της διαφθοράς και ε, στην κοινωνία αλλά και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Φυσικά θα μπορούσε να ε, βοηθηθεί ε, κατά αυτόν τον τρόπο ακόμα και η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε την έκθεση θα θέλαμε να αυξήσουμε ε, την προστασία και να ξέρουμε ποιες είναι οι υπάρχουσες εμπειρίες. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια ε, νόμιμη προστασία των καταγγελόντων από το 1963 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ε, πρέπει και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσπαθήσουν πραγματικά να εξασφαλίσουν την προστασία στο πλαίσιο αυτής της έγκαιρης προειδοποίησης, όπως κάνει το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, η Σλοβακία και πολλές άλλες χώρες. τις περισσότερες χώρες από αυτές βέβαια υπάρχει μια διαδικασία προειδοποίησης ε, μόνο εν μέρη και ε, είναι θεσμοθετημένοι σε διάφορους νόμους. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε τους εσωτερικούς μηχανισμούς ε, στο πλαίσιο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν χρησιμοποιούμε νομίζω ε, επαρκώς την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών, δηλαδή να εποφελούμαστε όλοι από τις καλύτερες πρακτικές που υπάρχουν σε άλλες χώρες. Εμείς, για παράδειγμα, στην Τσεχία έχουμε μία μερική προστασία και θα θέλαμε να θεσμοθετήσουμε κάπως διαφορετικά τα πράγματα, να υπάρξει ένας νέος νόμος. Πριν το κάνουμε αυτό όμως θα θέλαμε να ξέρουμε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Γι' αυτό εγώ θα προτείνω κάποιες τροπολογίες. Ε, δεν συμφωνούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια κοινή ε, νομική ε, διευθέτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Ντέτμαρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κρασνοντέμσκι για την παρουσίαση της ε, γνωμοδότησής του. Είναι επιτέλους καιρό, συμφωνούμε όλοι, για την νομική προστασία ε, των καταγγελόντων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο παρελθόν έχει πιέσει το Κοινοβούλιο πολύ την Επιτροπή, αλλά η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει νομοθετική πρόταση ακόμα, κάτι που για μένα είναι απολύτως απαράδεκτο. Αν οι καταγγέλλοντες ε, φτάσουν στο δικαστήριο να καταθέσουν ε, ε, για θέματα φοροαποφυγής ας πούμε που μπορεί κάποιες άλλες ε, κάποιες εταιρείες να κατηγορούνται πώς θα καταθέσουν χωρίς να υπάρχει προστασία είναι πολύ σημαντικό οι, οι πολύ σημαντικοί καταγγέλλοντες γιατί έτσι αποκαλύπτεται κάθε παράνομη δραστηριότητα, παρατυπία είναι συνεπώς πολύ σημαντική για την προστασία ε, του ευρύτερου κοινού για την εξασφάλιση της διαφάνειας, ε, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της φοροαποφυγής. Και υπάρχουν ε, βέβαια και πάρα πολύ σημαντικές μεγάλες εταιρείες ε, που πρέπει και αυτές να συμφωνήσουν με τις κυβερνήσεις. Νομίζω ότι οι καταγγέλλοντες είναι ο καλύτερος τρόπος να μάθουμε πολύ σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να αποκαλυφθούν. Η προστασία λοιπόν των ανθρώπων αυτών είναι πάρα πολύ σημαντική ε, για ε, τον πλουραλισμό των απόψεων, τη δημοκρατία, την ελευθερία και πιστεύουμε ότι, όπως λέει και ο κύριος Κρανστονοντέμσκι, ότι πρέπει να προωθείτε και σε επίπεδο πολιτικής αγωγής, δηλαδή πρέπει να γίνει μια προσπάθεια εκπαίδευσης και κατάρτισης όσον αφορά την ευαισθητοποίηση. Θα ήθελα επίσης να πω ότι οι καταγγέλλοντες ε, ε, έχουν, διατρέχουν έναν επαγγελματικό και προσωπικό κίνδυνο πολλές φορές ε, αποκαλύπτοντας κάποιες πληροφορίες και πρέπει να σκεφτούμε τι είδους αντιστάθμιση ή αποζημίωση θα μπορούσε να υπάρχει για τους καταγγέλλοντες. Αναμένω εναγωνίως την καλή συνεργασία και ελπίζω ότι θα βρούμε μια ικανοποιητική ε, λύσεις στην προστασία των καταγγελόντων. Ε, τους ανθρώπους όπως ο Ραφαέλα λέει και Αντουάν Ντετούρ θα μπορούν να καλύπτονται από τέτοιου είδους νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μίχελς για την ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε όσον αφορά την αντιμετώπιση των καταγγελτών ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα ήθελα να σε πιστήσω την προσοχή σε ένα βασικό πρόβλημα το οποίο ανακύπτει σχέση με αυτή την έκθεση. Ο εισηγητής ήδη ευθύ εξ αρχής λέει ότι οι πολιτιστικές διαφορές όσον αφορά την αντιμετώπιση των καταγγελτών στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπαρκτές και γι' αυτό το λόγο μεταξύ άλλων οι μηχανισμοί προστασίας οι μηχανισμοί προστασία τους θα πρέπει να ρυθμίζονται καλύτερα σε εθνικό επίπεδο. Πολιτιστικές ιδιαιτερότητες υπάρχουν φυσικά, αυτή είναι η αλήθεια. Εάν θέλουμε να δούμε τη γερμανική μετάφραση δεν έχουμε καν ένα σωστό όρο. Ε, αυτός ο οποίος δίνει κάποιες επισημάνσεις ε, ε, λέγεται στα γερμανικά. Ε, χωρίς τις πολιτιστικές ε, ιδιαιτερότητες ε, βεβαίως ε, θα πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δημοσιοποιούν ε, εγκλήματα τα οποία διαπράττονται εκ μέρου των τραπεζών ε, ή των οικονομικών συμφερόντων διώκονται και διακυβεύεται η ίδια η ζωή τους. Ο Αντουάν Ντεβέλτ παράδειγμα. Όσον αφορά τώρα τους δημοσιογράφους εδώ δεν χρειάζεται να γίνει καμία επισήμανση στις πολιτιστικές διαφορές. Η Επίτροπος λέει ότι ο Τέτερ και ο Χαλιέ έκαναν πραγματικά το σωστό, ότι πρόκειται για ένα ηθικό ζήτημα δεν ε, πρόκειται εδώ για πολιτιστικές διαφορές. Ως πολιτικοί που ασχολούμεθα με τα ζητήματα του πολιτισμού θα πρέπει να ε, μεριμνήσουμε για την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα των πολιτών να υπάρξει επαρκής διαφώτιση εκεί όπου αποτυγχάνουν οι κρατικές ε, δομές Ούτε Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξουν ενωσιακοί μηχανισμοί ε, προστασίας για αυτούς που αποκαλύπτουν αυτά τα μυστικά. Υπό την έννοια αυτή θα υποβάλουμε εμείς τις δικές μας τροπολογίες και χαίρομαι για την ε, συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Εύαντς. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα ζήτημα ε, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για μας και επηρεάζει βέβαια όλους τους τομείς ε, και βέβαια το θέμα του εκπαίδευση και του πολιτισμού που μας απασχολεί εμά αυτή την Επιτροπή. Είναι σημαντικό να υπάρχει λοιπόν νομική ασφάλεια, ασφάλεια δικαίου, νομική προστασία για τους ανθρώπους αυτούς και νομίζω ότι αυτό που θέλουμε είναι ένα κοινό ελάχιστο επίπεδο προστασίας ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι πολίτε να μπορούν να ασκούν αυτό το θεμελιώδε δικαίωμά του, ε, να ορθώνουν το ανάστημά τους ε, έναντι στην κακοδιαχείριση ή στα κακό κείμενα. Ε, βέβαια πρέπει να προωθήσουμε και μια κουλτούρα λογοδοσίας και ακαιρεότητας στο δημόσιο τομέα αλλά και στον ιδιωτικό τομέα και νομίζω ότι μπορεί να ε, βοηθήσει και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών που αυτό είναι κάτι που γνωρίζουμε χρειάζεται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή η κοινωνία. Ε, θα έπρεπε να υπάρχουν εσωτερικές διαδικασίες αλλά και εξωτερικές δίωδοι προκειμένου οι καταγγέλλοντε να μπορούν να καταγγείλουν κάτι στα μέσα ενημέρωση, σε μη κυβερνητικού οργανισμούς. Ε, ε, θα έπρεπε να μπορούν να υποστηρίζονται στο να αναλαμβάνουν δράση με κάθε προστασία βέβαια σε αντίπεινα, γιατί αυτό θα το κάνουν για το κοινό καλό. Δεν ξέρουμε κατά πόσο βέβαια, σαφώς πρέπει να υπάρχει μια προστασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όμως θα έπρεπε να ε, μην ε, παρεμποδίζονται κάποια κράτη-μέλη να επιφέρουν ακόμη με υψηλότερο επίπεδο προστασίας από το κοινό, αν το επιθυμούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ε, κύριε Κραστοντέμσκι, και εμείς θα υποβάλουμε τροπολογίες εκ μέρους της ομάδας μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω την εργασία του κυρίου Κάσνοντεύσκη σε σχέση με το ότι λαμβάνουμε υπόψη τις πολιτισμικές δυσκολίες που έχουν ε, μεγάλη επίπτωση στο περιβάλλον της πληροφορίας. Ο καταγγέλων προβαίνει σε μία πράξη ευθύνης και γι' αυτό θα πρέπει να τύχει προστασίας και στις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις προτεραιότητες των κρατών μελών, έχει σημασία να υπάρχει ε, και ένα είδος διδασκαλίας ε, για τους καταγγέλλοντες. Εμείς ε, έχουμε εντάξει αυτά τα στοιχεία, κυρίως προστασίας Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και τα συναφή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, θα ήθελα να παρακαλέσω την Επιτροπή να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα θέλαμε να πούμε καταρχήν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σημερίζεται το στόχο προστασίας των καταγγελόντων δημοσίου συμφέροντος και τον Ιούλιο του 2016 τόνισε ότι θα προβεί σε οριζόντιες ή τομεακές ε, δράσεις με βάση την αρχή της επικουρικότητας για την προστασία των καταγγελόντων. Υφίσταται ήδη κάποια μορφή προστασίας ε, στην ε, τομεακή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το πρόγραμμα εργασίας του 2017 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 3 ε, Μαρτίου μέχρι και τις 29 ε, Μαΐου έχουμε κινήσει μια διαδικασία διαβούλευσης και αυτή τη στιγμή γίνεται μια μελέτη αντικτύπου. Τα αποτελέσματα θα είναι έτοιμα στις αρχές Ιουνίου. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά της έρευνας θα προβούμε σε περαιτέρω δράσεις εκεί όπου χρειάζεται. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελες να πεις πάλι κάτι εκ μέρους του εισηγητού, ολοκληρώνοντας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ε, παρατήρησα ότι υπάρχει ένα εύρος ε, συζήτηση σε σχέση με τις πολιτιστικές διαφορές που ε, συνδέεται περισσότερο με τις εκπαιδευτικές διαδικασίες εντός των χωρών παρά τις ε, διαφορετικές ρυθμίσεις στην κάθε χώρα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια επαρκής κατάρτιση και αναμένω με ενδιαφέρον το τι θα, πώς θα αποφανθούν οι διάφορες επιτροπές επί του θέματος αυτού. Ευχαριστώ πολύ και μια παρατήρηση από τη δική μου πλευρά προς την Επιτροπή την Κομισιόν. Νομίζω ότι όλοι επισημάναμε ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι, ούτως ώστε οι δημοσιογράφοι, αλλά και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι προβαίνουν σε αποκαλύψεις, να προστατεύονται παρκώς εφόσον και ε, βεβαίως ε, θα πρέπει να τράσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ίσως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου ούτω ώστε να περάσουμε σε συγκεκριμένες ε, πράξεις. Γιατί ε, πολλοί καταγγέλλοντες αυτή τη στιγμή είναι εκτεθειμένοι. Άρα θα πρέπει να βρεθεί μια ευρωπαϊκή λύση ούτως ε, ώστε να εξασφαλίζεται παρκώς η προστασία των πηγών αλλά και οι καταγγέλλοντες να προστατεύονται εφόσον ε, εργάζονται προς το δημόσιο συμφέρον. Και εδώ δεν θα πρέπει να χάσουμε περισσότερο χρόνο η έκθεση της Νομικής Επιτροπής το καθιστά επίσης ε, σαφές και η δική μας δομοδότηση άλλωστε, άλλωστε βασίζεται σε αυτή τη γενική διαπίστωση. Η προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών είναι 29 Μαρτίου στις 6 ε, το απόγευμα και η ψηφοφορία στην Επιτροπή έχει προβλεφθεί για τις 30 Μαΐου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα διεξαχθεί τον Ιούνιο αυτού του έτους. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ και Τώρα θα περάσουμε στην ακρόαση εν σχέση με την μελέτη πίζα. Αλλά έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ίσως ε, μπορούμε να κάνουμε μια παύση μέχρι τις ε, δεκάμιση. <laughs>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

Thank Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε κάπως λιγότεροι, πάντοτε συμβαίνει αυτό μετά τις πάσει. Παρ' όλα αυτά ελπίζω να έρθουν κάποιοι συνάδελφοι, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντική η συζήτηση εδώ που θα μας απασχολήσει για δύο ώρες, τις επόμενες δύο ώρες. Θα ασχοληθούμε με τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα της ε, μελέτης ΠΙΖΕ. Το πρόγραμμα αυτό είναι μια τριετή της ε, έρευνα η οποία θέλει να αξιολογήσει εκπαιδευτικά θέματα ελέγχοντας τις δεξιότητες και τις γνώσεις των μαθητών. Για τις ευρωπαϊκές χώρες η μελέτη αυτή είναι μια σημαντική πηγή πληροφόρησης και για το στρατηγικό πλαίσιο της ε, Ευρωπαϊκής, ε, της, του θεματολογίου Ευρώπη 2020 και για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ακριβέστερα είναι η βάση για το benchmark ε, όσον αφορά τις ε, γνώσεις των 15χρονων ε, μαθητών. Το, όσον, στους τομείς και των μαθηματικών. Και θα πρέπει το κομμάτι των αδύνατων μαθητών να είναι κάτι του 15%. Ε, ελέγχθηκαν ε, οι περισσότερες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δημοσιεύθηκαν στις 6 Δεκεμβρίου του 2016 και μετά τα πρώτα πορίσματα οι χώρες μέλη δείχνουν μια μεγάλη διακύμανση όσον αφορά το κομμάτι των αδύναμων μαθητών στα μαθήματα αυτά. Για να τους βοηθήσουμε λοιπόν και για να κατανοήσουμε καλύτερα τα αποτελέσματα και να δούμε τι θα πρέπει να γίνει στο μέλλον, έχουμε πέντε ομιλητές εδώ, τους οποίους θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά και θα ήθελα να τους παρουσιάσω συντομία. Είναι ο Γιούρι Μπελφάλη, επικεφαλής του τμήματος Early Childhood and Schools ε, ε, μετά ο Γιάν Πακούλσκι ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Άντρης επικεφαλής της σχολικής επιθόρησης στην Τσεχία ο Γιώζεφ Πάζλ επικεφαλής της ε, μονάδα στο τμήμα της επιθεωρήσεων από την επιθεώρηση των τσεχικών σχολείων της Τσεχίας, η Πέτρα Φόκτ από το τοπικό κοινοβούλιο του North Rhine-Westfalen και εκπρόσωπος της Τσεντεού για την εκπαιδευτική πολιτική στο τοπικό κοινοβούλιο και ο Χωσέ Χουστίνο, ε, πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και πρώην Υπουργός Εκπαίδευσης στην Πορτογαλία. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω όλους που ήρθατε εδώ, αλλά πριν δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μου, επιτρέψατε μου δύο παρατηρήσεις. Ε, δεν είναι κακή ε, βούληση όταν σας εγκαταλείψω εδώ, ε, αλλά θα πρέπει να φύγω και η συνάδελφος κυρία Πόσκο θα αναλάβει το συντονισμό της συζήτησης. Επίσης θα ήθελα να δώσω το λόγο αν συντομία στην κυρία Σάντοβα η οποία ήταν, είχε πάρει την πρωτοβουλία για τη σημερινή συνεδρίαση και είχε προτείνει να ασχοληθούμε με τα απορίσματα της μελέτης αυτής και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως στο πλαίσιο της Επιτροπής μας στη συνεδρία των συντονιστών εγκρίναμε αυτή την πρόταση με μεγάλη μας ευχαρίστηση. Γι' αυτό θα ήθελα να της δώσω το λόγο για πέντε λεπτά. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε εδώ τους προσκεκλημένους μας. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία, γιατί μπορούμε να ε, συζητήσουμε τους, ε, τα αποτελέσματα των υπολογισμών μας ε, για το πίζα του 2015 και να κάνουμε και μία σωστή αξιολόγηση των συστημάτων εκπαίδευσης. Κάθε τρία χρόνια, όπως είπες Πέτρα, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τα αποτελέσματα των μαθητών, των σπουδαστών μας. Θέλουμε να είμαστε καλύτεροι, όμως βλέπουμε ότι συχνά έχουμε προβλήματα. Δεν βελτιωνόμαστε βελτιωνόμαστε. Δεν βελτιωνόμαστε. Ε, τα αποτελέσματα του ΠΙΣΑ ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά σήμερα ως δείκτης ε, και αν θέλουμε να επιτύχουμε υψηλή απασχολησιμότητα, πρέπει να, να, κοιτάμε τη βαθμολογία, γιατί δείχνει, δείχνει την απασχολησιμότητα, απασχολησιμότητα και την τα αποτελέσματα ε, στο σχολείο και όπως επίσης να δούμε και το θέμα πώς συσχετίζεται με την εγκατάλειψη του σχολείου. Ε, περίπου το 12% ε, των 12χρονων δεν επιτυγχάνουν ένα επαρκές επίπεδο εκπαίδευσης. Για μας λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία. Η κατάσταση αυτή γεννάει πολλά ερωτηματικά και πολλές προκλήσεις ε, σε κάθε επίπεδο, σε επίπεδο ε, όσα, σε επίπεδο κρατών μελών, σε επίπεδο σπουδαστών. Υπάρχουν μεθοδολογικές αλλαγές που έχουν γίνει στα κράτη-μέλη και αυτό είναι μία ερώτηση προς τον ε, συνάδελφο από το, στον προσκεκλημένο από τον ΩΣΑ πώς συσχετίζονται αυτά τα πράγματα, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα αποτελέσματα για τη βελτίωση του σχολικού συστήματος και την αποφυγή της ανεργίας. Η, το τρέχον επίπεδο συνεργασίας ε, ΩΣΑ και Ευρωπαϊκή Ένωσης είναι παρκές. Ελπίζω ότι η ακρόαση αυτή θα μπορέσει να βοηθήσει στην εξέβρεση απαντήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν τους μας και με χαρά θα ακούσω τις παρουσιάσεις τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σόντροβα, για αυτή τη σύντομη παρουσίαση και θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω τους ομιλ... θα πέρασω τώρα στους ομιλητές μας. Έχουμε χωρίσει την ακρόαση σε δύο τμήματα. Το ένα τμήμα, στο πρώτο τμήμα θα μιλήσουν ο κύριος Μπελφάλη και ο κύριος Πακούλσκι και στη συνέχεια θα ακολουθήσει γύρω ερωτήσεων και απαντήσεων και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο τμήμα του πάνελ και θα δώσουμε ε, το λόγο στους υπόλοιπους ομιλητές. Ε, κύριε Πελφάλη, σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Έχετε το... Ε, κυρία Πελφάλη, έχετε το λόγο. Ε, Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ γιατί ε, θέλετε να ε, μιλήσουμε για την απόδοση των ε, μαθητών και συναφή ζητήματα μέσω της διαδικασίας της πίζας. Μέχρι πέρσι το Δεκέμβριο φτάσαμε στα συμπεράσματά μας με βάση τη διαδικασία της πίζας και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βελτιώσουμε τα εκπαιδευτικά συστήματα παντού. Η Μιχαέλα σας είπε ότι η πίζα είναι ένα μέσον έτσι ώστε οι χώρες να ξέρουν πού βρίσκονται σε σχέση με τις επιδόσεις των μαθητών. Όχι μόνο ακαδημαϊκά, αλλά και πώς τα καταφέρνουν ως προς τη ε, ζωή μέσα στο σχολείο και εκτός αυτού, καθώς και τα κίνητρα μάθησης. Αυτό μας δίνει πολλές πληροφορίες για να κατανοήσουμε τι θα μπορούσαν να κάνουν περαιτέρω οι χώρες για να βελτιώσουν την ε, ποιότητα της εκπαίδευσης. Θα σας δώσω λοιπόν ορισμένα στοιχεία ως προς τις ε, ε, διεθνείς πρόπτικες και θα ακούσω και άλλους συνοδέλφους που θα μιλήσουν περισσότερο για τις ευρωπαϊκές ε, πρόπτικες και τις συναφείς συζητήσει. Το 2015 η Πίζα κάλυπτε 70 χώρες. Δεν πρόκειται για χώρες του ΩΣΑ μόνο, αλλά χώρες του ΟΣΑ και άλλες χώρες εταίρους και έχουμε περισσότερες χώρες που προσχωρούν. Θα έχουμε 80 χώρες το 2017 ε, και πιστεύουμε ότι θα είναι ένα διεθνές μέσον για να μπορέσουμε να έχουμε συγκριτικά στοιχεία για τις ε, επιδόσεις των μαθητών. Με βάση ε, το, τη διαδικασία της πίζας το 2015 μιλήσαμε για επιστημονική γνώση δηλαδή το πώς οι μαθητές μπορούν να ασχοληθούν με θέματα ε, που άπτονται της επιστήμης. Θέλουμε λοιπόν να δούμε πώς ε, αφομοιώνουν οι μαθητές την επιστημονική γνώση σε σχέση με τη φυσική, χημεία και ούτω καθεξής και πώς μπορούν να εγκολποθούν αυτά τα ε, δεδομένα, να μπορούν να ε, λύνουν και ζητήματα, προβλήματα ή θεωρίες και πώς μπορούν να σκέφτονται ως επιστήμονες για να αντιμετωπίσουν τα θέματα που θα τους απασχολήσουν στην ε, ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία αργότερα. Αυτό είναι ένα από τα μαθήματα και παραδείγματα. Άρα, ε, μιλάμε και για συγκεκριμένα, συγκεκριμένες δοκιμασίες με βάση ε, στοιχεία, στοιχεία ε, με τον υπολογιστή για να μπορούν να απαντούν σε επιστημονικά ζητήματα. Δηλαδή, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς μπορούν να μπορούν τα διάφορα σχήματα ή υποθέσεις και να προτείνουν απαντήσεις. Αυτό περιλαμβάνει ε, δοκιμασίες ε, κατανόησης του περιεχομένου αλλά και της επιστημονικής διαδικασίας για να δώσουν απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Εάν δείτε τα γενικά αποτελέσματα των γνώσεων, των επιστημονικών γνώσεων με βάση τη διαδικασία της πίζας, ε, λάβαμε υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα και ότι ακριβώς μέσα στα πλαίσια της ε, διαδικασίας ε, απόκτησης επιστημονικών γνώσεων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κινητή τηλεφωνία, τα κινητά, οι ταμπλέτες, το διαδίκτυο βοήθησαν αυτή τη διαδικασία. Ε, μιλάμε για μία ε, διαδικασία ε, επιδόσεων. Αρχικά βλέπετε ένα 400-450 και με βάση την ε, ψηφιοποίηση και τους αναπτυξιακούς στόχους τεχνολογίας μπόρεσαν να κατανοήσουν καλύτερα τις διαδικασίες αυτοματισμού ή την εξοικονόμηση ενέργειας όπως το αυτόματο αυτοκίνητο αλλά η κατάσταση του επιστημονικού αλφαβητισμού δεν έχει αλλάξει άρδιν. Βλέπετε ε, εδώ τι γίνεται στην ε, βιοχημία, στην ε, τρισδιάστατη ε, τεχνολογία, έτσι ώστε να υπάρχει ένα καλύτερο γνωστικό περιεχόμενο. Μεταξύ αυτών των χωρών είδαμε και χώρες που καταβάλουν προσπάθειες να βελτιώσουν τις συνολικές επιδόσεις των μαθητών. Όπως στην περίπτωση της Πορτογαλίας. Η Πορτογαλία έδειξε μία συνεχή βελτίωση ε, ως προς το γνωστικό περιεχόμενο και η Σιγκαπούρη που ήταν ήδη καλή ε, έφτασε σε επίπεδα αριστείας. Άρα το ζήτημα είναι να δούμε τι κάνουν αυτές οι χώρες για να βελτιώσουν αυτό το πλαίσιο και πώς οι άλλες χώρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να υποβοηθήσουν αυτή την ε, γνωστική διαδικασία η πίζα δεν αφορά μόνο ένα γενικότερο βαθμολόγιο, αλλά έχει σημασία να φτάσουμε σε μία εξισορρόπηση μεταξύ της ε, ποιότητας της εκπαίδευσης και της ε, ισομερούς ε, κατανομής της διαδικασίας. Βλέπετε δεξιά χώρες που τα καταφέρνουν και στην ποιότητα και στην ε, ίση πρόσβαση. Δηλαδή, άλλες βρίσκονται σε επίπεδο πάνω από αυτό του μέσου όρου του, του ΩΣΑ και αυτό σημαίνει ότι οι χώρες αυτές δημιουργούν και την θέληση στους μαθητές έτσι ώστε να μην λάβατε υπόψη μόνο το οικονομικό υπόβαθρο, οικογενειακό υπόβαθρο των μαθητών. Έτσι αυτοί οι μαθητές μπορούν να έχουν υψηλότερες επιδόσεις, βλέπετε. Ορισμένες χώρες όπως την ε, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Εσθονία, Φιλανδία όπου συνδέουν και τους δύο παράγοντες την ποιότητα και την ίση πρόσβαση, την ισότητα. Και βλέπετε και τις χώρες που προσπαθούν να προωθήσουν και τους ε, δύο τομείς, ε, και την ποιότητα και την ίση πρόσβαση. Και εάν δείτε τις ε, διαφορές επιδόσεων μέσα στην ίδια χώρα, μπορείτε να έχετε πολύ σημαντικά ευρήματα, δηλαδή τη διαφορά μαθητών από ένα φτωχό περιβάλλον και τους άλλους μαθητές, ας πούμε, στην ε, δημοκρατία του Δομήνικου, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ φτωχών και πλουσίων. Βλέπετε λοιπόν αυτό το διαχωρισμό, δηλαδή τα κόκκινα στίγματα σας δείχνουν ποιες είναι οι επιδόσεις των μαθητών από ένα μη προνομιακό περιβάλλον. Βλέπουμε επίσης ότι το, το μέγεθος του χάσματος είναι διαφορετικό μεταξύ χωρών. Δηλαδή, μερικές χώρες έχουν υψηλότερο χάσμα σε σχέση με τα προηγούμενα αποτελέσματα με βάση τη διαδικασία της πίζας και βλέπουμε ότι η φτώχεια δεν αποτελεί πεπρωμένο. Γιατί βλέπουμε ότι πολλοί μαθητές που ε, προέρχονται από ένα μη προνομιακό περιβάλλον τα καταλαβαίνουν πολύ καλά. Βλέπουμε την Εσθονία, Βιετνάμ, ε, Κίνα δηλαδή ε, μαθητές που προέρχονται από ένα πολύ φτωχό οικογενειακό περιβάλλον έχουν τις ίδιες επιδόσεις με άλλους. Με το μέσο όρο δηλαδή του όσα. Και υπάρχουν και χώρες που θέλουν να μειώσουν αυτή τις χαμηλές επιδόσεις και αυτή η γραφική παράσταση σας δείχνει ότι μπορούμε να προωθήσουμε αυτούς τους στόχους και να μειώσουμε τις χαμηλές επιδόσεις, το μερίδιο των χαμηλών επιδόσεων, γιατί υπάρχουν χώρες όπου οι μαθητές ε, μπορούν να ανταποκριθούν. Υπάρχει ένα ε, θα μπορούσαμε να πούμε πρόσημο ανθεκτικότητας, δηλαδή προερχόμενοι μαθητές από ένα φτωχό ή οικογενειακό περιβάλλον μπορούν να ανταποκριθούν στα κριτήρια της πίζας. Και αυτό το βλέπουμε και ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή η Εστονία έχει ευρωπαικες χωρες δηλαδη η Εσθονία εχει μαθητες που προέρχονται από ένα χαμηλό οικονομικό κοινωνικό περιβάλλον αλλά έχουν πολύ υψηλές επιδόσεις. Ως προς τις ε, καλύτερες επιδόσεις βλέπετε εδώ τον επιμερισμό των κρατών. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε μέσα στην ίδια χώρα ποια είναι η ποσοστιαία αναλογία των ε, μαθητών που βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο και το οποίο σημαίνει ότι αυτό από εδώ προέρχονται και οι μελλοντικοί επιστήμονες και μηχανική. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και παγκόσμια ποια, ποιος είναι ο καταμερισμός. Δηλαδή και στις ΗΠΑ βλέπουμε ότι οι υψηλές επιδόσεις δεν είναι τόσο υψηλές πραγματικά, αλλά επειδή πρόκειται για μεγάλη πληθυσμιακή κατηγορία φαίνονται περισσότερο. Η Ιαπωνία τα καταφέρνει πολύ καλά και ως προς το μέγεθος της χώρας και ως προς τις υψηλές επιδόσεις. Γι' αυτό και έχουν, κατέχουν μεγάλο μέρος, μεγάλο μερίδιο της πίτας. Ενώ στην Ευρώπη βλέπουμε ότι μέσα στην ίδια χώρα μπορούν να υπάρχουν υψηλές ή χαμηλότερες επιδόσεις, ανάλογα με τη χώρα. Μιλάμε για ένα 23% σε σχέση με το παγκόσμιο μερίδιο υψηλών επιδόσεων. Η πίζα δεν αφορά μόνο τις επιδόσεις, όπως βλέπουμε σήμερα, αλλά ρωτούμε τους μαθητές εάν θέλουν να ε, ασχοληθούν με την επιστήμη της επιστήμης όταν ενηλικιωθούν. Ορισμένες χώρες έχουν πολύ καλές επιδόσεις όπως η Γερμανία, η Φιλανδία. Αλλά αυτοί που θέλουν να μπουν, να, να μπουν στον θετικό τομέα έχουν πολύ μικρό μερίδιο. Ενώ αντίθετα βλέπουμε ότι σε άλλες χώρες, ενώ οι υψηλές επιδόσεις δεν είναι πραγματικά υψηλές, υπάρχουν μαθητές οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με τις επιστήμες. Θέλουμε λοιπόν να ε, προωθήσουμε τους μαθητές προς αυτή την κατεύθυνση έτσι ώστε να ασχοληθούν με αυτές τις ε, προκλητικές ε, με επιστήμες που παρουσιάζουν μεγάλες προκλήσεις. Θα πρέπει να κατανοήσουμε επίσης ότι οι επιδόσεις σχετίζονται και με τη χαρά της γνώσης καθεαυτή. Άρα για τα εκπαιδευτικά συστήματα, στα εκπαιδευτικά συστήματα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όχι μόνο τις υψηλές επιδόσεις, ένα σύστημα επιδόσεων καθαρά, αλλά να προωθήσουμε και την θέληση μάθησης. Και αυτό ιδιαίτερα στον επιστημονικό τομέα. Άρα, για να ε, έχετε χρόνο και για συζητήσεις. Θα χρησιμοποιήσω μόνο τις ε, δύο τελευταίες διαφάνειες. Δεν μιλάμε μόνο λοιπόν για βαθμολόγια εδώ και για επιδόσεις, αλλά και το κατά πόσο οι μαθητές θέλουν να χρησιμοποιήσουν την ε, επιστήμη στην καθημερινή του ζωή και πώς θέλουν να έχουν μια επιστημονική σταδιοδρομία. Βλέπουμε ορισμένες χώρες που πληρούν τα δύο και τα τρία κριτήρια, μεταξύ των οποίων και ορισμένες ε, ευρωπαϊκές χώρες. Μπορείτε λοιπόν να διαβάσετε την έκθεσή μου και θα ήθελα να πω ότι η πίζα κινείται πέρα από θέματα επιστημονικού αλφαβητισμού. Οι χώρες προσπαθούν να λάβουν υπόψη τις ε, ε, αρμοδιότητες, ε, τις επιδόσεις, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να ανταποκριθεί. Πώς, μπορεί, πώς μπορούν οι μαθητές να ανταποκριθούν και στα επιστημονικά δεδομένα στην καθημερινή τους διαβίωση. αυτοί που αποφασίζουν θέλουν να δουν πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ε, ε, μαθητές να ε, ζουν καλύτερα σε μία διαφοροποιημένη κοινωνία. Δηλαδή, παραμένοντας την ίδια τους στη χώρα, θα πρέπει να μπορούν να διαδράσουν και με ανθρώπους που προέρχονται από ένα διαφορετικό πολιτισμικό ή γλωσσικό περιβάλλον. Και να ανταποκριθούν και στα ζητήματα της κοινωνίας. έτσι ώστε να μπορέσουν να εργαστούν επικοδημητικά για την ευημερία ολόκληρη της κοινωνίας. Άρα θα ήθελα να γίνουν συζητήσεις για το ποιες αρμοδιότητες, ποιες επιδόσεις θα πρέπει να μας απασχολήσουν για το μέλλον μέσα στα πλαίσια των μελλοντικών επιδόσεων και βαθμολογίου της πίζας. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ε, επισκόπηση. Ε, ξέρω πόσο δύσκολο είναι μέσα σε 10 λεπτά να παρουσιάσει κανείς πραγματικά τα πολύ ε, λεπτομερή αποτελέσματα αυτής της μελέτης, αλλά νομίζω μας δώσετε μια πολύ καλή εικόνα ε, για τα αποτελέσματα της μελέτης και πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Πακούλσκι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας παρουσιάσει τις δικές του αξιολογήσεις σε σχέση με την έρευνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε σε αυτή τη σημαντική συνεδρίαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, και την κυρία Σοντοβα, η οποία ε, ήταν υπεύθυνη για την ε, οργάνωση. Θα ήθελα επίσης ε, να σας πω ότι εμείς θέλουμε να διευκολύνουμε μια ενημερωμένη συζήτηση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον εκπαιδευτικό τομέα. Δεν είναι γνωστό γεγονός, αλλά από τον περασμένο Νοέμβριο περάσαμε σε μια άνευ προηγουμένου περίοδο, στην οποία θα έχουμε πρόσβαση σε άνευ προηγουμένου ε, δεδομένα τα οποία αφορούν τον εκπαιδευτικό τομέα από διάφορες πηγές. Η πίζα είναι ένας, ε, μία από αυτές τις πηγές, όπως είπε και συνάδελφος προηγουμένως. Ε, αυτό έχει άμεση σχέση με έναν από τους έξι πίνακες επιδόσεών μας για την χαμηλή επίδοση. Δεύτερον, φέτος χαιρόμαστε ιδιαίτερως γιατί για πρώτη φορά όλα τα κράτη-μέλη έχουν συμμετάσχει σε αυτήν την έρευνα, οπότε αυτό μας δίνει πολύ πλούσιο υλικό, ε, το οποίο είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε πλήρως. Αυτές οι δύο παρουσιάσεις ε, ταιριάζουν πολύ γιατί προφανώς ο σα είναι ο πρώτος ε, οργανισμός που ε, είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των δεδομένων αυτών ε, και συμπεριλαμβάνει και χώρες που είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως. Εμείς επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι συστάσεις πολιτικής έχουν άμεση σχέση με τα πορίσματα. Θα τα ακούσετε λοιπόν και από μένα. Θα υπάρχουν φαντάζομαι και αντίτυπα στην αίθουσα. Θα αρχίσουμε όμως από την προηγούμενη πίζα του 2012 όταν συνεργαζόμενοι με τον ΩΣΑ πριν από την ε, αποκάλυψη των αποτελεσμάτων συνεργαστήκαμε πάρα πολύ για τις συστάσεις πολιτικών ε, που προκύπτουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση από την έρευνα αυτή. διαθέσαμε, τα διαθέσαμε στην, ε, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αυτό νομίζω ότι μιλά από μόνο του όσον αφορά την ε, ύπαρξη μιας ενημερωμένης συζήτηση ε, για την κατάσταση των 15χρονων μαθητών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, Ξεκινώντας θα έλεγα ότι για μας αυτό ε, αποτελεί ένα είδος αφύπνισης γιατί αν πάμε πίσω στο 2009 μετά στο 2012 πιστεύαμε πολύ ότι η Ευρώπη ήταν στο σωστό δρόμο, δεν πήγαινε πολύ γρήγορα αλλά τουλάχιστον πήγαινε προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα πιο πρόσφατα ε, συμπεράσματα αποτελέσματα δεν το δείχνουν ε, όμως αυτό. Αυτό είναι μια κακή έκπληξη και πρέπει να μας ε, ε, αφυπνήσει λιγάκι, ειδικότερα ως προς τις επιστήμες. Όπως βλέπετε, και η συνάδελφος το ανέφερε προηγουμένως, ε, ε βλέπετε πως είναι η κατάσταση, είναι αρκετά ε, αξιοσημείωτη στις επιστήμες. Να δούμε επίσης και ξεχωριστά κάποιες χώρες. Αυτό ε, είναι ενδιαφέρον αν δει κανεί ότι το 2012 είχαμε τέσσερις χώρες ε, που ανταποκρίνονταν στο ε, benchmark μετά ήταν μόνο τρεις οι χώρες, οι περισσότερες χώρες δηλαδή πήγαν προς τα πίσω. Ε, περιέργως η Πορτογαλία και η Σουηδία κατάφεραν να πάνε αντίθετα στο ρεύμα και σημείωσαν βελτίωση και ε, η δημοσίευσή μας ε, δίνει ιδιαίτερη σημασία στο ποιο ήταν το μυστικό πίσω από τις επιδόσεις αυτών των δύο χωρών. στο, στην επόμενη γραφική παράσταση βλέπετε ακριβώς τις διαφορές, μία μεθοδολογική παρατήρηση, γιατί μπορεί κάποιοι να εκπλαγείται από τις δύο παρουσιάσεις ο όσα χρησιμοποιεί μη σταθμισμένους μέσους όρους. Εμείς ε, περιμένουμε βέβαια να, βλέπουμε, δούμε την ε, ε, επίδοση της συνολική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το βαθμολογικό πίνακα επιδόσεων όσα επικεντρώνεται περισσότερο σε επίπεδο κρατών μελών, βλέπετε ότι οι ανισότητες, οι διαφορές είναι μεγάλες μεταξύ των ε, ε, χωρών. Συγγνώμη, έχω ξεχάσει τα γυαλιά μου και δεν μπορώ να δω ε, ακριβώς σε ποια διαφάνεια είστε. Δεν, δεν μπορείτε να μου το δείξετε σε μια πιο κοντινή οθόνη. Όχι. Ε, τότε αν κάνω λάθος ε, θα με συγχωρέσετε. Όσον αφορά τώρα τις ε, συστάσεις ε, για τις πολιτικές, αυτό αντλεί από τα διδάγματα της δικής μας ανάλυσης. Έχουμε, θεωρούμε ότι Πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης ε, με, μέσω της επένδυσης και στην αρχική αλλά και στη συνεχή ε, κατάρτιση των διδασκόντων. Η διαχείριση των σχολείων επίσης είναι πολύ σημαντικά. Ε, η προσέγγιση του συνολικού σχολείου είναι επίσης κάτι που μας φαίνεται ενδιαφέρον. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τώρα ε, άλλους τομείς, είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση όσον αφορά την ανάγνωση σε σχέση με τη διαφορά μεταξύ των δύο φύλων θα δείτε ότι για κάποιες χώρες, ότι, θα δείτε ότι για κάποιες χώρες η διαφορά είναι πολύ σημαντική. Αυτή η διαφάνεια δείχνει πώς ε, έχει εξελιχθεί η διαφορά μεταξύ των φύλων μεταξύ του 2012 και του 2015. Μειώνεται το φάσμα, αλλά όχι αρκετά γρήγορα. Και ενδιαφέρον είναι ε, σε σχέση με τα αποτελέσματα από τους ε, ομοτήμους που καλύπτουν δηλαδή και, άλλα, και άλλες ηλικιακές ομάδες, μειώνεται αυτό το, το, χάσμα. τα αγόρια βελτιώνονται σε σχέση με τα κορίτσια, όμως δεν αλλάζει το γεγονός ότι εξακολουθούν να έχουν χειρότερες επιδόσεις. Ε, βλέπετε πολύ συγκεκριμένες συστάσεις και εδώ δεν χρειάζεται να τις ε, διαβάσω. Πάντως είναι ε, πορίσματα του, της Γενικής Διευθυνσής μου ε, και, υπάρχει και το, και υπάρχουν και οι βέλτιστες πρακτικές που ακολούθησαν τα κράτη-μέλη. Κάτι ακόμη πολύ σημαντικό για μας είναι οι επιδόσεις ε, όσων έχουν χαμηλότερες επιδόσεις. Ε, στις επιστήμες είναι η χειρότερη κατάσταση. Η Εσθονία είναι η μόνη χώρα η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή ακριβώς στο, στο, στο, στο σημείο το σωστό του βαθμολογικού πίνακα ε, και ε, τα μεγαλύτερα προβλήματα σημειώνονται στα πιο μειονεκτούντα άτομα ε, που δεν είναι πλήρως ενταγμένα. Ε, επικεντρωνόμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό τους μαθητέ χαμηλών επιδόσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας δείχνω πόσο μεγάλε μπορεί να είναι οι διαφορές μεταξύ των αντίστοιχων χωρών και θα ήθελα να ε, σας ε, παροτρύνω να δείτε ε, ποιες είναι οι πολιτικές που προτείνουμε να αναλάβουν, να ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη. Οι επιδόσεις των μεταναστών μας ενδιαφέρουν πολύ για προφανείς λόγους. Τα κράτη-μέλη κάνουν πολύ σημαντικές προσπάθειες να εντάξουν τους μετανάστες. Ε, θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να ρίξετε, να, να, ρίξετε μια ματιά ε, στις λεπτομέρειες, στα λεπτομερή στοιχεία που έχουμε για την ομάδα αυτή. Πάλι είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Κάποιες ε, συστάσεις προκύπτουν επίσης. Ε, συνεργαζόμαστε και πολύ στενά με τη Eurostat ε, για να μπορούμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα δεδομένα για τις μεταναστευτικές ροές. Μία ακόμη διάσταση είναι το ζήτημα το, της, της απόδοσης του εκπαιδευτικού συστήματος και βλέπουμε ότι οι χώρες που επενδύουν ε, στην ε, προσχολική ηλικία και στην εκπαίδευση προσχολική ηλικία τα καταφέρνουν καλύτερα και αυτό είναι κάτι που ε, πρέπει να το επισημαίνουμε πάντοτε όταν μιλάμε για τις επιδόσεις των 15χρονων παιδιών. Θα ήθελα λοιπόν αυτά σε γενικές γραμμές να σας αναφέρω για να βοηθήσω τη συζήτηση. Τη συζήτηση. Εμείς έχουμε τρεις σημαντικές ε, εκθέσεις αυτή τη στιγμή. Μία από κοινού με τον ΩΣΑ που αφορά ειδικότερα το θέμα της, ε, των, επιδόσεων ε, των 15χρονων μεταναστών. Επίσης περιμένουμε τα αποτελέσματα δύο ακόμη μελετών. Μία αφορά τους μετανάστες και την γλωσσική πτυχή της ένταξής τους και μία ακόμη, η οποία επίσης μπορεί να είναι πολύ διαφωτιστική είναι ποια είναι τα μυστικά πίσω από τον περιορισμένο αριθμό πολύ καλών ε, επιδόσεων ε, ατόμων με πολύ ε, φτωχό, με πολύ φτωχή προέλευση. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά ήταν αυτά που ήθελα να σας πω. Θα περιμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βακούλσκι. Τώρα έχουμε χρόνο για ορισμένες ερωτήσεις ή παρεμβάσεις. Η κυρία Σάντροβα έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Έχω δύο ερωτήσεις. Χαιρετίζω την, ε, ε, την ε, συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον ΩΣΑ. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή απόφαση ε, και όσον αφορά την μεθοδολογία και την ε, οικονομική υποστήριξη. Ίσως θα μπορούσατε να σχολιάσετε το εξής. Έχετε το στόχο να γίνει η μελέτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετάσχουν όλες οι χώρες. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας πολύ θετικός στόχος. Και έχω και μια ερώτηση στον κύριο Πακούλσκι. Δεν ήξερα πώς, δεν, ξέρω πώς οι ευρωπαϊκές ε, χώρες μπορούν να μοιραστούν τις βαλίστες πρακτικές. Βεβαίως μπορούν ε, να συναντηθούν όπως ε, για παράδειγμα στο Ελσίνσκι υπάρχουν ορισμένες συνεδριάσεις ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνετε κάποια ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ανάπτυξη των συστημάτων αξιολόγησης, της εκπαίδευση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Για την κυρία Γιούρη θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πώς χρησιμοποιείτε ως όσα τα αποτελέσματα ε, της μελέτης σας ε, σε άλλες μελέτες για διατύπωση συστάσεων προς άλλες ε, χώρες. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που εδώ έχουμε μία... Ε, σήμερα έχουμε μία διερμηνία από τα σλοβενικά και μπορώ να μιλήσω σλοβενικά. στην ε, εκπαιδευτική διαδικασία υπάρχουν διαφορές μεταξύ των φύλων. Και διαπιστώνουμε επίσης ότι υπάρχουν άλλοι παράγοντες που καθορίζουν τη σχολική επιτυχία. Ωστόσο, βλέποντας αυτά τα αποτελέσματα, και αυτό αφορά κυρίως τη δυνατότητα ανάγνωσης, διαπιστώνουμε ότι τα κορίτσια είναι πολύ καλύτερα από τα αγόρια. Και διερωτώμε λοιπόν πού παρατηρούνται οι διαφορές αυτές ε, μεταξύ των δύο φύλων. Γιατί εγώ ε, πιστεύω βεβαίως τα κορίτσια είναι πιο πετυχημένα από τα γόρια. Όχι μόνο στις βασικές γνώσεις όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες, αλλά αργότερα στο Λύκειο. Ε, πώς εμφανίζεται αυτή η διαφορά μεταξύ των φύλων. Παρακαλώ και τους δύο μιλητές να μου δώσουν μια απάντηση. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ριμπέρο θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα χρησιμοποιήσω τη δυνατότητα να μιλήσω πορτογαλικά. Ε, εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης, όχι της Επιτροπής Πολιτισμού. Παρ' όλα αυτά, το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την απασχόληση στην Ευρώπη. Εγώ είμαι καθηγήτρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ε, ασχολούμαι ε, με όλα όσα αφορούν τους καθηγητές. Η Πίζα θέλει να, δει, να κοιτάξει προς το μέλλον. Έχω το εξής ερώτημα όσον αφορά τις ειδικότητες. Θα ήθελα να γνωρίζω, θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο μπορείτε να μου πείτε πώς ε, είναι δυνατόν να αποκτηθούν ε, όλες αυτές τις σφαιρικές γνώσεις τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη γιατί μελλοντικά θα αυτοματοποιηθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας και οι νέοι άνθρωποι βρίσκονται έναντι μια τεράστια πρόκληση. Θα πρέπει να ασχοληθούν με τα ρομπότ, με την τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Αυτό θα είναι καθοριστικό στοιχείο για την απασχόληση. Και διερωτώ κατά πόσο εμείς δεν θα έπρεπε να κινηθούμε στην κατεύθυνση αυτή ούτως ώστε οι νέοι άνθρωποι να αποκτήσουν και αυτές τις δεξιότητες. Ευχαριστούμε. Κύριε ναι, Χέγκοφ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω την εξής ερώτηση. Πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε τις ε, ήπιες ε, δεξιότητες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ειδικοτήτων. Γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν επαγγέλματα της, ε, στο πλαίσιο της επαγγελματικής ε, εκπαίδευσης, τα οποία μπορούν να αξιολογηθούν ε, εύκολα. Αλλά πώς θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε τις λεγόμενες ήπιες δεξιότητες που δεν είναι στο πλαίσιο της επίσημης εκπαίδευσης. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα έχουμε την κυρία Χέλγα Τρούπελ και στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε τις απαντήσεις. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της αφεκτικότητας ορισμένων μαθητών, γιατί είπατε ότι 25% πραγματικά έχουν πολύ καλές επιδόσεις, έστω και αν προέρχονται από φτωχό περιβάλλον ε, κοινωνικά και οικονομικά. Ε, είναι ένα θέμα νοημοσύνης. Ε, τι είναι αυτό που τους προσδίδει αυτή την ικανότητα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια πληθώρα ερωτήσεων και θα μπορούσατε να συμφωνήσετε ποιος από τους δύο θα ξεκινήσει. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Ο κύριος Πακούλσκι. Ευχαριστώ. Θα αλλάξουμε ε, μεταξύ μας και θα, κάπως θα διαχωρίσουμε τις ερωτήσεις. Η δική μας ε, ε, συνεργασία ε, έχει ενισχυθεί, υπάρχουν διεθνείς συναντήσεις κορυφής ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ΟΣΑ. Ε, και σημαντικούς φορείς εκπαίδευσης. Υπάρχει ένα ολόκληρο πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο αναπτύξαμε μαζί με τους συναδέλφους του αρμοδίου τμήματος του ΟΣΑ και εχουν επενθει επενδυθεί 2-3,5 εκατομμύρια ευρώ σε αυτή τη συνεργασία. Όσον αφορά τη συμμετοχή στις ε, διεθνείς ε, μελέτες, ε, νομίζω ότι η στάση είναι πολύ θετική. Υπάρχουν όλο και περισσότερες χώρες που συμμετέχουν στις μελέτες. Η Πίζα βεβαίως είναι μια ακραία περίπτωση ε, θα θέλουμε να υπάρξει πιο μεγάλη εκπροσώπηση, πιο μεγάλη συμμετοχή. Υπάρχει βεβαίως ένα θέμα του κόστος και μια κόποση. Ε, προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτά τα θέματα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι το εξής. Ε, η ανταλλαγή βελτιστών πρακτικών. Θα πρέπει να πω ότι από τη δική μας προεπτική εμείς ε, παρακολουθούμε συστήματα εκπαιδευτικής ε, κατάρτισης. Όσον αφορά τα benchmarks και τις ε, ενδείξεις, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν και εισφέρουν, συνεισφέρουν παράχον, παρέχοντας δεδομένα. Επίσης υπάρχουν και ομάδες εργασίας που είναι μια άλλη δυνατότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω με την ευκαιρία αυτή την Ολλανδική Προεδρία γιατί κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας ε, έγινε μια συνεδρίαση ε, σε σχέση με τα στοιχεία που μπορούμε να έχουμε για την ε, βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Υπάρχουν πολλές μελέτες που τρέχουν και θα έχουμε πραγματικά μια πληθώρα δεδομένων και αυτό μας δίνει μια σημαντική ευκαιρία, σημαντικές ευκαιρίες για να αυξήσουμε τις γνώσεις μας στο τομέα αυτό προκειμένου να προβούμε σε μια ανταλλαγή βαλτίστων πρακτικών μεταξύ των χωρών μελών. Ίσως ε, η Γιούρη θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Γιάννη. Το θέμα του κατά πόσο οι χώρε μπορούν να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα τη ΠΙΖΑ ε, για την χάραξη των πολιτικών του και πώ μπορεί να συσφιχθεί η συνεργασία, θα ήθελα να πω ότι ήδη συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κάνουμε μια εισβάθος ανάλυση των δεδομένων τη μελέτη ΠΙΖΑ. Ε, Το Δεκέμβριο είχαμε τα αδρά αποτελέσματα, αλλά θέλουμε να συνεργαστούμε ώστε να, γίνουμε, να γίνει μια ε, ανάλυση κατά θεματολογικούς τομείς ο ΣΑ κατόπιν αιτήματος των χωρών προσπαθεί να προχωρήσει σε μια σβάθα ανάλυση των αποτελεσμάτων και κατανάλυση στα αποτελέσματα υπό το πρίσμα των ε, πολιτικών, των εκπαιδευτικών πολιτικών των διαφόρων χωρών μελών. Για παράδειγμα, ε, με την ε, Τσεχία ζητήματα ισότητας ή στην Σουηδία ε, έγινε η προσπάθεια να γίνει μια ανάλυση ε, των αποτελεσμάτων και της φθήνουσας ε, πορείας, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα τα αποτελέσματα. Έχουμε λοιπόν κάποιες δυνατότητες ε, συγκεκριμένης συνεργασίας με επιμέρους χώρες. Όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, ε, ε, στην επευκαιρία της Διεθνούς ημέρας των γυναικών προβάλαμε τα αποτελέσματα, αλλά το θέμα αυτό αφορά κυρίως την ανάγνωση, αλλά όχι τα μαθηματικά, γιατί εκεί τα αγόρια είναι πολύ καλύτερα από τα κορίτσια. Αλλά αν δείτε τις χαμηλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς, διαπιστώνετε ότι υπάρχουν περισσότερα αγόρια παρά κορίτσια όσον αφορά τις χαμηλές επιδόσεις. Αλλά αν δούμε και τις ε, top επιδόσεις, εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν περισσότερα αγόρια παρά κορίτσια. Εκεί το μερίδιο των κοριτσιών είναι ισχνότερο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το καταλάβουμε εις βάθος το θέμα αυτό όσον αφορά τον διαχωρισμό των δύο φύλων, αλλά και επίσης τα κίνητρα που υπάρχουν από πίσω, γιατί τα κορίτσια παρόλο που κινούνται στο ίδιο επίπεδο επιδόσεων με τα αγόρια, έχουν λιγότερη εμπιστοσύνη όσον αφορά τα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης ε, τα μαθηματικά για παράδειγμα έχουν περισσότερο άγχος και δεν αισθάνονται παρκώς προετοιμασμένα για καριέρες ε, στα σταδιοδρομή μαθηματικών. Άρα λοιπόν ε, ένα ρόλο παίζει επίσης και οι προσδοκίες των γονέων καθώς και η στάση των καθηγητών. Τέλος, ορισμένοι συμμετέχοντες έφτιαν το θέμα του πώς μπορούμε να μπούμε σε νέους τομείς όπως είναι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, να δούμε πού βρίσκονται οι διάφορες ε, χώρες και ποιες δυνατότητες υπάρχουν απόκριση αντίδρασης σε θέματα, για παράδειγμα, τεχνητής ε, νοημοσύνης. Αναγνωρίζουμε τη σημασία του να κατανοήσουμε ε, πού βρίσκονται οι διάφορες χώρες στον τομέα αυτό. Αλλά δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό οι μαθητές ε, αποδεικνύουν την ικανότητα, έχουν την ικανότητα να ζήσουν σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό ε, σε, στην κάθε χώρα οι μαθητές είναι εξοπλισμένοι με την ικανότητα, έχουν την ικανότητα να συνεργαστούν με άλλους. Γι' αυτό προσπαθούμε στο επίπεδο του ΟΣΑ να κάνουμε ένα διεθνές benchmarking. Είναι δύσκολο να γίνει συγκρίση μεταξύ των χωρών. Προσπαθούμε όμως να ορίσουμε τομείς όπου είναι δυνατόν να γίνουν συγκρίσεις επί τη βάση ξεκάθαρων ορισμών αυτού του οποίου θέλουμε να αξιολογήσουμε, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ιδιομορφίες της κάθε χώρας. Το 2015 κάναμε μια μελέτη επαλήθευσης η οποία δείχνει ότι τα τεστ πίζα ε, ε, μπορούν να συμπεριλάβουν τις δεξιότητες επικοινωνίας των ε, μαθητών. Αλλά υπό το πρίσμα της προόδου της επιστήμης ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε με δύο τρόπους. Το ένα είναι τι δεξιότητε θα πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές ούτω ώστε να μπορούν να εργάζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και να μπορούν να υποφεληθούν ε, βεβαίως από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Αλλά το άλλο κομμάτι αυτής της τόσο σημαντικής συζήτησης είναι το πώς θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε την ε, συμβολή των ανθρώπινων όντων τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι εδώ, ούτω ώστε η δική τους εισφορά να είναι όλο και πιο σημαντική. Μιλάμε για την ε, σημασία της δημιουργικότητας. Θα πρέπει ε, λοιπόν να εξελίξουμε ε, δεξιότητες τις οποίες δεν μπορούν ε, να εκτελέσουν τα ρομπότ η δυνατότητα της ενέστησης, η δυνατότητα της ε, δημιουργικότητας. Ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία για να απειλήσουμε θέματα όμως τα οποία μπορούν να προωθήσουν μόνο τα ανθρώπινα όντα και όχι υπολογιστές αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και την ευρωπαϊκή οπτική εδώ. Τι ακριβώς εσείς συζητάτε με πολιτικούς όρους. Για να επεκταθώ στα σχόλια του Γιούρη, ως προς τα δύο φύλλα, στα θέματα παγκόσμιας αρμοδιότητας, όπως είπε και η Γιούρη, έχει μεγάλη σημασία να σταθούμε στις βασικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίστηκαν μερικά χρόνια πριν. Θα πρέπει να μας απασχολήσουν απόλυτα μέσα στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εξελίξεων και μία συνολική αποτίμηση σε τεχνικό επίπεδο και επίπεδο πολιτικών για να δούμε ποιες είναι οι βασικές αρμοδιότητες. Αυτό σχετίζεται και με το benchmarking που προανέφερε ο συνάδελφος ε, δηλαδή το πλαίσιο του 2020 αποτελεί μία διαδικασία που μας ε, οδηγεί σε μια διαδικασία οριοθετήσεων. Μιλάμε για έξι οριοθετήσεις, έξι benchmarks. Τώρα θα μπούμε στο έβδομο και αυτό που είναι σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσουμε πλήρως τα περισσινά δεδομένα και να δούμε πώς ε, μπορούν αυτά τα benchmarks να μας βοηθήσουν στα κράτη-μέλη. Υπ' αυτή την έννοια θα πρέπει να μας απασχολήσουν οι βασικές ε, αρμοδιότητες σε θέματα οριοθέτησης. Δεν μπορούμε να έχουμε πολλά ε, ε, πληθώρα δηλαδή benchmark γιατί τότε χάνουμε το στόχο μας. και σε σχέση με τα στοιχεία που ορίζουμε προς τα κάτω, έχει σημασία η μέτρηση, η καταμέτρησή τους και η επικοινωνία. Βρισκόμαστε σε ένα πρώτο στάδιο τεχνικού επίπεδου. Αυτό που έχει σημασία είναι να φτάσουμε σημασία έχει να δώσουμε σημασία στις προκλήσεις για να δούμε πώς θα καλύψουμε τις ήπιες δεξιότητες. Θα ήθελα λοιπόν να λάβουμε ε, υπόψη μεθοδολογικά στοιχεία τα οποία θα ορίσουν και την πορεία μας. Να απαντήσετε και στο θέμα της ανθεκτικότητας. Είπατε ποιος είναι ο λόγος ε, πίσω από αυτή την ανθεκτικότητα. Από ό,τι βλέπουμε στα στατιστικά στοιχεία, αυτό που έχει σημασία είναι η κατανομή των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή, ποια είναι η κατανομή πόρων στα σχολεία που μειονεκτούν γιατί πολλές φορές τα σχολεία που πλεονεκτούν είναι αυτά που έχουν και περισσότερους πόρους. Και αυτό που έχει σημασία είναι ε, οι μαθητές που μειονεκτούν να τύχουν μεγαλύτερης υποστήριξης. Σε ορισμένες ε, χώρες οι δάσκαλοι, οι καθηγητές πάνε στα σχολεία που έχουν διοριστεί και λογοδοτούν με βάση αυτό το σύστημα αξιολόγησης της χώρας. Αλλά ορισμένες χώρες ενθαρρύνουν τους καθηγητές στην συνεργασία για να βοηθήσουν τους μαθητές που μειονεκτούν. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι να ε, υποστηρίξουν οι καθηγητές, να υποστηρίζονται, ιδιαίτερα σε σχέση με τους ε, μαθητές που μειονεκτούν. Θεωρούμε δηλαδή ότι τα θέματα ανθεκτικότητας και επιμονής μπορούν να λυθούν κατάλληλα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη, το πρώτο πολύ ενδιαφέροντα γύρο. Και τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο τμήμα της ανταλλαγής ε, Πάψαν και θα ήθελα να δώσω το λόγο στους δύο Τσέχους συναδέλφους, ο κύριος Ανδρέη Άντρης και ο κύριος Γιώσεφ Πάσελ, ε, πέντε λεπτά έκαστος. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. θα μιλήσω γαλλικά αυτή τη φορά και θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα την κυρία Μιχαέλα Σόιδρεβα γιατί μας κάλεσε για να σας μιλήσουμε για την ε, πείρα μας και τις εμπειρίες μας με βάση το μηχανισμό της πίζας στην τσεχική δημοκρατία. Θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω τον φορέα μας που είναι υπεύθυνο για την πραγματοποίηση, για την υλοποίηση των στόχων της πίζας. Η γενική επιθεώρηση εκπαίδευσης έχει ήδη συσταθεί το 18ο αιώνα σε, στην εποχή της Μαρίας Θηρεσίας και επιβίωσε μέχρι σήμερα. Πρόκειται για μια εθνική αρχή που δημιουργήθηκε με νομοθέτημα και που βοηθά το Υπουργείο Εθνικής Εκπαίδευσης έτσι ώστε να βοηθήσουμε για την ποιότητα της εκπαίδευσης, της δημόσιας εκπαίδευσης στα σχολεία. Η γενική, γενική επιθεώρηση εκπαίδευσης της τσεχικής δημοκρατίας βρά σε επίπεδο κράτους και μας απασχολεί και η διεθνή συνεργασία, δηλαδή πολλές δραστηριότητες για, την, ε, για τις ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίσης μέσα στα πλαίσια του Εθνικού Κέντρου Ερευνών η Εθνική Επιθεώρηση Εκπαίδευσης προσπαθεί να προβάλλει ε, μία, ε, μία εθνική συγγνώμη, διάσκεψη επιθεωρητών που είναι πολύ γνωστή στην Ευρώπη. Είμαστε υπεύθυνοι σε πολλούς τομείς αξιολόγησης των ε, συνθήκων εκπαίδευσης καθώς και των επιδόσεων των μαθητών. Πρόκειται για τρία, τρεις τομείς που, είναι, που αλληλοσυμπληρώνονται. Δεν μπορούμε να κρίνουμε την ποιότητα χωρίς να επιβλέπουμε το εκπαιδευτικό σύστημα. Και επίσης ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το εκπαιδευτικό γίγνεσθε και τα αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να κρίνουμε την ποιότητα όλων των σχολείων στη τσεχική δημοκρατία, καθώς και ολόκληρο το, σύστημα, ε, το εθνικό σύστημα εκπαίδευσης. Και όπως σας είπα, είμαστε υπεύθυνοι και για την υλοποίηση των ε, διεθνών ερευνών με βάση τη διαδικασία της πίζας. Στην τσεχική δημοκρατία Ακολουθούμε μία σειρά κριτηρίων και συνθήκων για να κρίνουμε τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Πρόκειται για ε, ένα πρότυπο που χρησιμοποιούμε, ποιοτικό πρότυπο, με βάση έξι κριτήρια. Το πρώτο αφορά την πλαισίωση του σχολείου, μετά ε, την ε, παιδαγωγική ηγεσία, την ε, ποιότητα του προσωπικού, του διδακτικού προσωπικού. Το τέταρτο ακολουθεί την εκπαιδευτική διαδικασία. Στη συνέχεια με τα αποτελέσματα και τέλος ο τελευταίος τομής είναι τα κριτήρια που αφορούν την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση. Κάθε κριτήριο εκπροσωπεί και αποτελεί μία περιγραφή, αποτελείται από μία περιγραφή γιατί η Γενική Επιθεώρηση Εκπαίδευσης αξιολογεί τα σχολεία χρησιμοποιώντας τέσσερα επίπεδα αρχίσουμε από το άριστα, ικανοποιητικά, το επίπεδο σύμφωνα το οποίο χρειάζεται βελτίωση και το ανεπαρκές και την ανεπάρκεια. Έχουμε δύο βασικά καθήκοντα. Καταρχήν να αποτιμήσουμε την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των σχολείων και το δεύτερο αφορά την ε, αποτίμηση ολόκληρη του εκπαιδευτικού συστήματος. Έχουμε ε, δύο ή τρία έγγραφα. Μετά από κάθε επίσκεψη σε σχολείο συντάσσεται μία έκθεση της επιθεώρησης όπου περιγράφεται το, η εκπαιδευτική διαδικασία και τα αποτελέσματά της σε επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο κάθε χρόνο συντάσσουμε την ετήσια έκθεση που είναι ένα πολύ βασικό έγγραφο που συζητείται σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο γερουσίας για να δούμε την διδακτέα ύλη, θετικές επιστήμες, ε, μαθηματικά και ούτω καθεξής. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου. Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω για τις ε, συγκριτικές μελέτες, γιατί πάντα χρειαζόμαστε feedback. Μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για μια διαδικασία ανάδρασης. Λίγο πιο αργά σας παρακαλώ, λέει η Πρόεδρος, γιατί οι διερμήσει είναι αδύνατο να σας παρακολουθήσουν. Μέσα στα πλαίσια της σχολικής επιθεώρησης δίνουμε ε, feedback σε σχολικό επίπεδο, το οποίο σημαίνει ότι γίνεται μία εξωτερική και εσωτερική αξιολόγηση και πάλι πιο αργά. Συνεχώς επιταχύνεται. Αν θέλετε να σας παρακολουθούν, να μιλάτε πιο αργά. Αυτό σημαίνει ότι η σχολική επιθεώρηση κάνει μία αξιολόγηση και μετά γίνεται και μία αυτοαξιολόγηση από τα σχολεία. Μετά έχουμε το εκπαιδευτικό σύστημα, την αποτίμηση εκπαιδευτικού συστήματος. Γίνεται ένας εσωτερικός ε, έλεγχος και λαμβάνουμε υπόψη και τις ε, θεματικές ενότητες Και αυτό που μας ενδιαφέρει επίσης είναι να απαντήσουμε και σε διεθνείς συγκριτικές μελέτες όπως αυτή της πίζας. Υπάρχει δηλαδή μία συνέργεια εσωτερικού και εξωτερικού επίπεδου μέσα στα πλαίσια των συγκριτικών μελετών. Αυτό που έχει σημασία είναι οι διεθνείς συγκριτικές αξιολογήσεις να μας δώσουν στοιχεία μέσα στα πλαίσια του συλλογικού αυτού γίγνεσθε. Εμείς συμμετέχουμε σε ε, διεθνείς μελέτες από το 1995. Η τρέχουσα συμμετοχή αφορά ε, πίσω teams Τάλις και Πέλτ. Και αυτές είναι οι τέσσερις συμμετοχές μας και φυσικά ε, χαιρόμαστε και για την ε, συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία μας βοήθησε να ε, συμμετάσχουμε και στο ICLS. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή αυτή η συμμετοχή αν και ξέρουμε ότι η μακροχρόνια ο μακροχρόνιος προγραμματισμός δεν είναι πάντα εφικτός. Θέλουμε όμως να υπάρχει μια συλλογική αξιολόγηση, γιατί έτσι είναι πιο εύκολο να δούμε πού μπορούμε να ανταποκριθούμε και πού όχι. Μιλάμε λοιπόν για την πίσα και εδώ έχετε μία συγκεφαλαίωση των κύκλων και βλέπετε ότι και για τους τρεις τομές, τομείς εδώ, δηλαδή ανάγνωση μαθηματικά και επιστήμονες, μπορέσαμε να καλύψουμε τους τρεις μεγάλους κύκλους και ε, γίνεται αποτίμηση του κάθε τομέα ξεχωριστά. Πώς εξελίχθηκε η δική μας ιστορία. Εδώ βλέπουμε την ε, ανάγνωση, τα μαθηματικά και το μαύρο είναι οι επιστήμονες, οι επιστήμες, συγγνώμη. Εδώ βλέπετε ποιες ήταν οι επιδόσεις στους τρεις τομείς, στους τρεις βασικούς τομείς. Και βλέπουμε ότι οι μαθητές μας έχουν χαμηλότερες επιδόσεις με το πέρασμα του χρόνου. Εδώ έγιναν δύο μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στις επιδόσεις των μαθητών. Το 2000 έγινε μία μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και για τα σχολεία σημαίνει μεγαλύτερη οικονομική αυτονομία και το 2005 αυτονομήθηκαν πλήρως τα σχολεία έτσι ώστε να μπορέσουν να δράσουν ανάλογα με τα προγράμματά τους. ο γυμνασιάρχης και λυκιάρχης είναι υπεύθυνος για όλα τα οικονομικά συστήματα ε, θέματα διαπαιδαγώγησης, ακόμα και τα, τα κτηριακά κατασκευαστικά. Φυσικά τα οικονομικά είναι το μείζον ζήτημα που τους απασχολεί. Η μεταρρύθμιση δημόσιας διοίκησης ε, σήμαινε υποστήριξη των, ε, του διδακτικού προσωπικού και των ε, γυμνασιαρχών λυκιαρχών. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις ίσως κινήθηκαν πολύ γρήγορα και ίσως η δημόσια διοίκηση δεν ήταν έτοιμη καθόλου. Ας δούμε τι κάνουμε σε επίπεδο επιθεώρησης. αυτού αυτή η ανακεφαλαίωση σας δείχνει όλα τα επίπεδα, δηλαδή ακαδημαϊκούς ερευνητές, ε, βουλευτές, ΜΜΕ, γυμνασιάρχες, λυκιάρχες και διδακτικό προσωπικό. Μέχρι τώρα έχουμε αποτελέσματα και με βάση την PISA 2015. Αυτή τη στιγμή γίνεται μία δευτερογενής ανάλυση για να ασχοληθούμε με επιμέρους ζήτημα. Προσπαθούμε να έχουμε ε, στέρεα θεμέλια με βάση τη χρήση των ε, μελετών της πίζας και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η επιλεξιμότητα γιατί βασιζόμαστε στα στοιχεία της εθνικής επιθεώρησης που δείχνουν ότι η εκπαιδευτική επιλεξιμότητα υπάρχει και αυξάνεται δυστυχώς. Και αυτό θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να πείσουμε τους εκπαιδευτικούς φορείς ότι θα ευεργετηθεί η κοινωνία πολύ περισσότερο εάν υπάρχει κάποια ετερογένεια στην ε, σύνθεση των τάξεων σε σχέση με άλλες χώρες. Σας ευχαριστώ. vielen herzlichen Dank. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για το παράδειγμα αυτό που μας δώσατε, δηλαδή πώς ε, μια χώρα ε, αντιμετωπίζει τα αποτελέσματα της μελέτης. Θα ήθελα να με συγχωρέσετε που είμαι λίγο αυστηρή όσον αφορά το χρόνο ομιλία. αλλά νομίζω ότι είναι πιο δίκαιο να επιτρέψουμε να μιλήσουν και οι άλλοι ομιλητές και ίσως να μείνει και λίγος χρόνος για τη συζήτηση. Λυπάμαι λοιπόν αν δείχνω το σφυρί μου όταν υπερβαίνονται τα όρια, τα περιθώρια του χρόνου μιλίας. Τώρα θα ακούσουμε την Πέτρα Φόκτ από την Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία. Γνωρίζετε ότι στη Γερμανία η εκπαίδευση εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ομόσπονδων κρατηδίων και όχι της κεντρικής κυβέρνησης. Είναι σημαντικό λοιπόν μια εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης να μας μιλήσει για τα εκπαιδευτικά θέματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσω τα αποτελέσματα από την πλευρά μιας χώρας ε, μέλης. Ε, μέλους. Ε, η Πίζα είναι μια μελέτη που συγκρίνει τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα ε, και από την άλλη συγκρίνει εσωτερικά τα αποτελέσματα του κάθε ομόσπονδου κρατηδίου. Όπως είπατε, στη Γερμανία υπάρχουν διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα ανακρατήδιο. Η πίζα μας δεν είναι στοιχεία για τα ελλείμματα των σχολικών συστημάτων και η σύγκριση αυτή ε, τόσο διεθνώς και η σύγκριση αυτή, μάλλον ε, τη σύγκριση αυτή δεν ήθελαν να την κάνουν οι περισσότεροι ε, αρμόδιοι για τα εκπαιδευτικά θέματα στη Γερμανία γιατί ε, θεωρούσαν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα του κάθε κρατηδίου είναι το καλύτερο από τα άλλα. Υπάρχει μια τάση τώρα στη Γερμανία να υπάρξει μια ενοποίηση όσον αφορά τα τις εξετάσεις για το σχολικό απολυτήριο. Τα σχολεία ελέγχονται στη Γερμανία βάσει ποιοτικών κριτηρίων ε, και αξιολογείται η ποιότητα, κάτι το οποίο στο παρελθόν ήταν αδιανόητο για τη Γερμανία. Αυτό οδηγεί σε μια καλύτερη συγκρισιμότητα των σχολικών συστημάτων στη Γερμανία και δίνει τη δυνατότητα να βρίσκουμε κάποια διδάγματα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά ε, συστήματα και να τα μεταφέρουμε στα άλλα ομόσπονδα κρατήδια. Τώρα, συγκεκριμένα, τι έχει γίνει σε σχέση με τα αποτελέσματα της ΠΙΖΑ, μπορούμε να πούμε ότι έγινε η προσπάθεια, τα ελλείμματα όσον αφορά την ανάγνωση να καλυφθούν με μια ενίσχυση της προσχολικής αγωγής. Ε, σημαντικό ρόλο παίζει εδώ η ε, πρόθεση της γλώσσας. Παιδιά τα οποία δεν μπορούν γλωσσικά να παρακολουθήσουν τι γίνεται στο μάθημα. Και δεν πρόκειται μόνο για παιδιά μεταναστών, αλλά και για Γερμανούς, οι οποίοι έχουν γλωσσικά ελλείμματα ήδη πριν ξεκινήσουν το σχολείο. Γι' αυτό αρχίσαμε να αρφανώζουμε διάφορα προγράμματα, τα οποία είναι προϋπόθεση, ούτως ώστε να ξεχωρίσουμε τις προϋποθέσεις για μια επιτυχή συμμετοχή στο σχολικό σύστημα οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες των ε, μειονεκτούντων μαθητών στόχος είναι βεβαίως να αυξηθούν. Στη Γερμανία υπάρχει το εξή πρόβλημα. Στο παρελθόν ε, ε, πάρα πολλοί μαθητές έλειπαν από τα μαθήματα και αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι ότι ισχυρίζονται το γεγονό ότι παιδιά από καλύτερες ε, οικογένειε, από υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο έχουν τη δυνατότητα ελλείμματα στο σχολείο να τα επεξεργαστούν και να τα καλύψουν στο σπίτι ενώ παιδιά από φτωχό περιβάλλον δεν έχουν τι αντίστοιχε δυνατότητες. Άλλο ερώτημα είναι τα στερεότυπα των φύλων σε σχέση με τα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης και πώς μπορούν να ξεπεραστούν αυτά τα στερεότυπα. Ε, υπάρχουν προγράμματα ενίσχυσης των μαθητών προς όλα τους μαθητές και με δεδηλωμένο στόχο να ενδιαφερθούν τα κορίτσια για τα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης, γιατί εδώ υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Υπάρχουν επιμέρους προγράμματα όπου ε, σκεφτόμαστε κατά πόσο έχει, ίσως δεν θα είχε νόημα να διαχωριστούν τα φύλλα σε συγκεκριμένους τομείς γιατί όχι μόνο μειονεκτούν τα κορίτσια σε, ορισμένα, σε ορισμένους τομείς, αλλά πολύ συχνά και τα γόρια έχουν προβλήματα με το σχολικό σύστημα. Αυτά τα προγράμματα διαχωρισμού των δύο φύλων είναι αρκετά μεμονωμένα μέχρι στιγμής, αλλά ωστόσο προσπαθούμε να τα εξειδικεύσουμε σε σχέση με το φύλο και να προωθήσουμε χωριστά το κάθε φύλο. Τώρα, όσον αφορά την ψηφιοποίηση, το αναφέρατε ήδη, ε, λόγω του μόσπονδου συστήματος, μοσπονδιακού συστήματος δεν παρεμβαίνει η κεντρική κυβέρνηση αλλά η αρμόδια υπουργός πρότεινε ένα ψηφιακό σύμφωνο γιατί διαπίστωσε ότι υπάρχει μια υστέρηση εδώ ε, στη Γερμανία. Πρότεινε λοιπόν αυτό το σύμφωνο ψηφιακής ε, εκπαίδευσης, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν κάποια θέματα χρηματοδότηση μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και κυβερνήσεων των ομόσπονδων κρατηδίων, αλλά από το, και από το 2018 ε, θα τρέξει αυτό το πρόγραμμα για πέντε χρόνια, πέντε δις ε, ευρώ είναι ο προπολογισμό. Ακόμα βρίσκει στη φάση προγραμματισμού και το συζητούν και γίνονται κάποιοι προβληματισμοί για το πώς ε, θα μπορούσαν ε, οι νεαροί άνθρωποι να προετοιμαστούν ε, καλύτερα για το ψηφιακό μέλλον που τους περιμένει στην αγορά. όσον αφορά τον εξοπλισμό των σχολείων, εδώ είναι οι τοπικές αρχές, οι κοινωτικές αρχές αρμόδιες Άρα είναι πολύ δύσκολο να ε, περάσουν κάποιες προτάσεις. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα των δήμων και των κοινοτήτων. Τα σχολεία στη Γερμανία είναι περίπου 40.000 και θα έπρεπε βεβαίως να εξοπλιστούν ε, τεχνικά, αλλά όπως σας είπα υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες, ε, ταμπλέτες, υπολογιστές κλπ. Ωστόσο, αυτό είναι σημαντικό θέμα. Βέβαια, η τεχνική δεν είναι αυτό σκοπό. Η μάθηση με ηλεκτρονικά μέσα θα πρέπει να έχει και μια παιδαγωγική αξία. Η δημόσια συζήτηση πηγαίνει προ την κατεύθυνση του να πούμε ότι όλα αυτά είναι σημαντικά για το μέλλον, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορεί κανείς να τα εξηγήσει θαυμάσια με τον μαυροπίνακα και την κοιμωλία. Δεν θα πρέπει να γίνονται τα πάντα ψηφιακά. Ένας άλλος σημαντικός τομέας είναι η επαγγελματική κατάρτιση. Και εδώ θα λίγο με κάποια αιτήματα για αύξηση του ποσοστού των, της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Αυτό είναι σημαντικό. Από την άλλη, στη Γερμανία έχουμε ένα πολύ σημαντικό και πετυχημένο σύστημα διτής ε, επαγγελματικής εκπαίδευσης που είναι ε, εγγύηση για την οικονομική δύναμη της Γερμανίας και το οποίο το έχουμε εδώ και πολλά χρόνια, είναι σημαντικό και έχει σαν αποτέλεσμα, και αυτό το έδειξαν πολλέ μελέτε ε, να μειωθεί η ανεργία των νέων και επίσης είχε σαν αποτέλεσμα η Γερμανία να σταθεί στα πόδια της ε, ε, καλύτερα από άλλες χώρες τελευταία οικονομική κρίση, γιατί υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι που έχουν ε, πάρει αυτή την επαγγελματική κατάρτιση και οι οποίοι δεν ε, απολύθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης με το επιχείρημα ότι ακριβώς ήταν το προσωπικό των επιχειρήσεων το οποίο οι ίδιες οι επιχειρήσεις είχαν καταρτήσει πολύ καλά. Στη Γερμανία έχουμε ένα δεύτερο πολύ πετυχημένο σύστημα λοιπόν ε, ε, ε, και ε, και, αλλά υπάρχει τάση παρόλα αυτά στη Γερμανία όλο και περισσότεροι να θέλουν να πάνε στα πανεπιστήμια, να έχουν μια ακαδημαϊκή εκπαίδευση, άρα ίσως μειώνεται αυτό το κομμάτι της διτής επαγγελματικής εκπαίδευσης και αυτό μας ανησυχεί. Γιατί ε, στη Γερμανία δεν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ακαδημαϊκά πτυχία, οι οποίοι έχουν ε, ευκαιρίες στην ε, αγορά εργασίας, αλλά μάλλον αυτοί οι οποίοι ακολουθούν αυτό, παρακολουθούν αυτό το διτό σύστημα επαγγελματική κατάρτισης και τελικά έχουν περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης από ό,τι οι έχοντες ακαδημαϊκό πτυχίο. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να εξοπλίσουμε με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας της επαγγελματικές αυτές σχολές, ούτω ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ε, παράλληλα προς, το, την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Γιατί πραγματικά δίνουμε μεγάλη αξία σε αυτή τη δυνατότητα και αυτό συνάδει και με τα αποτελέσματα της πίζα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον επόμενο ομιλητή. Κύριο Ζουστινό. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω πορτογαλικά, μια και έχω αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω την πρόσκληση αυτή για να ε, μιλήσω. Θα προσπαθήσω να συγκεντρώσω ορισμένα στοιχεία προσπαθώντας να ορίσω μια γενικότερη πλαισίωση και τα διδάγματα τα οποία αντλήσαμε από την εργασία της Πίζας και από τα αποτελέσματα ε, με βάση τις ε, τάσεις που καταγράφονται από το 2000 και μετά. Θα πρέπει να μην, μπούμε, να μην δεχτούμε αυτή τη διχογνωμία του αν είμαστε καλοί ή κακοί μαθητές. Δηλαδή θα πρέπει να αντλήσουμε ε, διδάγματα χωρίς να θέλουμε να ε, προβάλλουμε μία μανιχαϊστική προσέγγιση του καλού ή κακού μαθητή. Αυτή ακριβώς την εικόνα βλέπετε και εδώ, γιατί δεν θέλουμε να είμαστε καλοί ή κακοί μαθητές. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά εδώ αναφέρομαι σε τρεις ε, χώρες σε σχέση με την Πορτογαλία και επειδή τα αποτελέσματα είναι γνωστά δεν θα ήθελα να χάσω χρόνο με την ανάλυση αυτή, αλλά <coughs> να δούμε σε τι συμπεράσματα μπορούμε να φτάσουμε με ε, βάση αυτή την ανάλυση. βλέπουμε ότι υπάρχει σύγκληση αποτελεσμάτων με το πέρασμα του χρόνου. Οι χειρότερες χώρες δεν είναι στην ίδια θέση, ενώ οι χώρες με τα καλύτερα αποτελέσματα ε, αντιμετωπίζουν ε, το πρόβλημα του να παραμείνουν καλοί. Υπάρχει λοιπόν ένα φαινόμενο σύγκλησης το οποίο πρέπει να γνωστοποιήσουμε γιατί αυτό που έχει σημασία είναι ότι η οικονομική σύγκληση πολλές φορές οδηγεί και στην εκπαιδευτική ε, σύγκληση. Η Πορτογαλία από το 2000 και μετά ασχολήθηκε πολύ με την εκπαίδευση αλλά λίγο με την οικονομία. Δηλαδή, οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα 15 τελευταία χρόνια έγιναν μέσα σε μία δυσχερή οικονομική κατάσταση ε, λιτότητας και έτσι οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις έπρεπε να γίνουν με πολύ πιο ισχυρές πεπιθήσεις γνωρίζοντας ότι η καλύτερη λύση δεν προωθείται με περισσότερους οικονομικούς πόρους πάντα. Δηλαδή μέσα στα πλαίσια οικονομικής λιτότητας έπρεπε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της ε, εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Ποιοι ήταν οι παράγοντες που μας βοήθησαν στο να φτάσουμε σε καλύτερα αποτελέσματα σύμφωνα με την πίζα, μη έχοντας ε, η οικονομική υποστήριξη. Εδώ βλέπετε αυτούς τους άξονες ανάλυσης. Ε, διάλεξα τα μαθηματικά ε, στα χ και στα Y ε βλέπουμε το κατακεφαλή ΑΕΠ. Βλέπετε ότι η Πορτογαλία δεν είχε αύξηση του, του κατακεφαλή ΑΕΠ μεταξύ 2000 και 2012. Δηλαδή η οικονομική μας ανάπτυξη ήταν σχεδόν μηδενική, όμως στον εκπαιδευτικό τομέα είχαμε καλές εξελίξεις κάτι το οποίο μας οδηγεί σε ορισμένα συμπεράσματα. Ποια ήταν τα αίτια αυτής της ε, βελτίωσης τη στιγμή που δεν υπήρχαν χρήματα, δεν υπήρχαν οικονομικοί πόροι. Το επόμενο γράφημα σας ε, εξηγεί τους διαφόρους τομείς που βοήθησαν. Βλέπετε λοιπόν εδώ Δυστυχώς δεν είχα χρόνο να σας ε, μεταφράσω αυτή τη διαφάνεια στα αγγλικά, αλλά ο παράγων που υποβοήθησε τη βελτίωση αυτή ήταν το γεγονός ότι λάβαμε ε, υπόψη τα σχολεία όπου υπήρχαν μαθητές με χαμηλές επιδόσεις, δηλαδή κάναμε μία στοχοθέτηση των σχολείων και έτσι βοηθήσαμε τα συγκεκριμένα σχολεία. Ε, βλέπουμε λοιπόν καλύτερα αποτελέσματα. Άρα η εξέλιξη μεταξύ 2000 και 2012 αλλά και 2015 με τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε καλύτερα σχολεία. Βλέπουμε ε, λοιπόν ότι λαμβάνοντας υπόψη τις χαμηλές επιδόσεις βοηθήσαμε τα σχολεία που είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Το δεύτερο σχετίζεται με τους καθηγητές. Σήμερα έχουμε καθηγητές με καλύτερα προσόντα, δηλαδή έχουν εξειδικευτεί, έχουν μία ειδίκευση. Τώρα οι καθηγητές πρέπει να σπουδάσουν για πέντε χρόνια με δύο χρόνια ειδίκευση και αν το συγκρίνετε με το 2000 είναι ένα σημαντικός ε, λόγος για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Πέρα από αυτό υπάρχουν περισσότερα κίνητρα από ό,τι στο παρελθόν. Επίσης η αυτονόμηση των σχολείων, ένας παράγων Και υπάρχουν και αρνητικοί παράγοντες, δηλαδή η σημασία του ΑΕΠ, του κατακεφαλή ΑΕΠ. Η ποιότητα, η κτηριακή ποιότητα και κατασκευή σχολείων. Αυτό που μπορέσαμε να αναγνωρίσουμε ήταν ότι οι καθηγητές κάνουν τη διαφορά έχουμε καλύτερους καθηγητές, άρα και καλύτερους μαθητές. Δηλαδή, ακριβώς επειδή ε, ειδικεύονται περισσότερο οι καθηγητές, μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών. Η τελευταία γραφική παράσταση δείχνει κάτι το ενδιαφέρον. ότι δηλαδή ο καλός συσχετισμός και σχέση καθηγητών μαθητών είναι ένας άρρηκτος σύνδεσμος αυτής της, σχέδης, της σχέσης αιτιόδους συνάφειας που δείχνει ότι τελικά οι μαθητές νιώθουν καλύτερα στα σχολεία γιατί έχουν και καλύτερους καθηγητές. Και αυτό οφείλεται στις ε, εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, σε διαρθρωτικούς παράγοντες και θα ήθελα να σας πω πώς φτάσαμε σε αυτά τα καλύτερα σχολεία με καλύτερους καθηγητές από το 2000 κάνουμε μία νέα ε, οργάνωση των σχολείων και τα, έργανο τα οργανώνουμε σε school clusters έτσι ώστε να έχουμε μία πολύ καλή διάρθρωση ε, μεταξύ σχολείων με βάση την ε, διδακτέα ύλη. Και υπάρχει και εξωτερική αξιολόγηση των σχολείων από τη Γενική Επιθεώρηση. Επίσης, άλλαξε η παραδοσιακή διαχείριση των σχολείων. Σήμερα υπάρχει μία διαχείριση όπου ενισχύεται ο παιδαγωγικός χαρακτήρας. Ως προς το διδακτικό προσωπικό, ήδη αναφέρθηκα σε αυτό αυτό που έχει σημασία είναι και η εξωτερική αξιολόγηση ε, με δοκιμασία στο τέλος κάθε σχολικής περίοδου. Είχαμε δύο ε, δοκιμασίες οι οποίες απορρίφθηκαν, αλλά στο... τώρα υπάρχουν, γίνονται εξετάσεις τον ένατο χρόνο και την, ε, τον δωδέκατο, δηλαδή στο ΜΠΑΚ στο απολυτήριο. Τέλος, ε, αντιμετωπίζουμε δύο προβλήματα που ελπίζουμε να επιλύσουμε κατά τα προσεχή χρόνια. Η Πορτογαλία ε, δυστυχώς παρουσιάζει μεγάλο ποσοστό μετεξεταστέων, ένα από τα υψηλότερα επίπεδα της Ευρώπης. Και τι γίνεται με αυτό το τρόπο αποκλείονται, αποκλείονται μία μερίδα μαθητών καταστρέφοντας το ανθρώπινο δυναμικό μας. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να προωθήσουμε μία ειδική εκπαιδευτική διεργασία για τα επόμενα χρόνια. Επίσης χρειάζεται αποκέντρωση των εκπαιδευτικών πολιτικών. γιατί δυστυχώς στην Πορτογαλία υπάρχει μεγάλος συγκεντρωτισμός στην διοίκηση των σχολείων. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε αυτά τα δύο μεγάλα βήματα μεταρρύθμισης. Δηλαδή μπορώ να πω ότι ήμασταν τυχεροί που δεν είχαμε χρήματα τελικά γιατί χρειάστηκε να κάνουμε την εκπαιδευτική μας μεταρρύθμιση εκ των ενόντων. Ευχαριστώ πολύ. Αφού ακούσαμε τις παρεμβάσεις, Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, αν θέλουν να κάνουν παρατηρήσεις. Ένα-δύο λεπτά παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές για τις ενδιαφέρουσες ομιλίες του. Ε, διαπιστώνω πόσο σημαντική είναι η πίζα, ούτε ώστε επί τη βάση των αποτελεσμάτων να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών μελών. Μία ερώτηση σε σχέση με το διτό εκπαιδευτικό σύστημα οι περισσότερες χώρες επιθυμούν ε, να ε, εντάξουν στοιχεία του διτού εκπαιδευτικού συστήματος στη Γερμανία, γιατί στη Γερμανία τα αποτελέσματα είναι θαυμάσια. Ιδίως όσον αφορά τη μετάβαση από το σχολείο στο επάγγελμα. Και όπως είπαμε υπάρχουν χαμηλά ποσοστά αναργίας, αλλά είπατε ότι υπάρχουν και δυσκολίες μετά το, αυτό το διτό σύστημα εκπαίδευσης να ξεκινήσει κανείς ακαδημαϊκές σπουδές. Τι γίνεται με αυτό. Γιατί θα ήθελα να παρακολουθήσω τις εξελίξεις στη Γερμανία. Ευχαριστούμε και πάλι την κυρία Σοντρόβα για την πολύ καλή πρωτοβουλία διοργάνωσης αυτής της συζήτησης. Ευχαριστώ η κυρία Σοντρόβα. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο μιλήσω τσεχικά εφόσον έχω τη δυνατότητα για να θέσω κάποια ερωτήματα. Αυτό που με ενδιαφέρει ε, είναι η κατάσταση στη Γερμανία. Έχουμε τα αποτελέσματα πίζα της Γερμανίας και ομολογώ ότι δεν ξέρω πώς γίνεται η πίζα στην Γερμανία αν υπάρχει ένας οργανισμός που οργανώνει τις εξετάσεις σε ολόκληρη τη χώρα ή κάθε κρατήδιο οργανώνει ε, με το δικό του τρόπο το ε, πίζα. Ε, αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Επίσης, ε, κατόπιν των αποτελεσμάτων ε, της ΠΙΖΑ, είτε σε επίπεδο κρατηδίου, είτε σε επίπεδο ομόσπονδης Γερμανίας, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπήρξαν αντιδράσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι τον, ε, συνά, τον συνάδελφο τον Πορτογάλο, επειδή είπε ότι παρά τις δαπάνες για την εκπαίδευση, οι δαπάνες αυτές ακόμη και αν δεν έχει διατηρηθεί το ποσοστό ε, ε, ε, το, το, ποσοστό δαπανών προς την εκπαίδευση εξακολουθούν να υφίστανται βελτιώσεις στην, στις επιδόσεις και κατά πόσο πιστεύετε ότι η ποιότητα των σχολείων μειώνει ε, το ε, ποσοστό των μαθητών που έχουν χαμηλές επιδόσεις. Προφανώς ε, αυξήθηκαν οι πόροι προς, τους προς τα σχολεία. Ποια θα ήταν όμως μια διαφορετική μέθοδος προκειμένου να επιτύχουμε την ίδια βελτίωση. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση στην Τσεχία, πρέπει να πω ότι Λίγες είναι οι πιθανότητε να έχουμε πολιτική σταθερότητα. Εδώ και 10 χρόνια ε, έχουμε ήδη τον 10ο Υπουργό Παιδείας και η κατάσταση κάπως έχει σταθεροποιηθεί σήμερα. Αυτό μπορεί να έχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Πιστεύω όμως ότι ε, μία από τις πτυχές που δεν αξιολογήθηκε ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε από τον ΩΣΑ ε, που προσθέτει, συνεισφέρει στην ε, βελτίωση της ποιότητας είναι η πολιτική σταθερότητα. Να υπάρχει μια συνέχεια όσον αφορά τις πολιτικές, ε, τις εκπαιδευτικές. Χωρίς πολιτική σταθερότητα αμφισβητούνται τα αποτελέσματα και ε, θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσει ο συνάδελφος από την Τσεχία. Όσον αφορά τώρα την αποκέντρωση και τη σχετική παρατήρηση για την Πορτογαλία, θα ακούσατε αυτό που υπόθηκε από τον κύριο Βασού. Το σύστημα ε, είναι πολύ αποκεντρωμένο στην Τσεχία και αυτό έχει βέβαια ως αποτέλεσμα και κάποιες κινδύνους. Πολύ καλή είναι η αποκέντρωση, αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Μήπως υπάρχει κανείς άλλος που θέλει να πάρει το λόγο ενώ όχι, να ξαναδώσω ε, το λόγο στους εμπειρογνώμονές μας για να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω με το ερώτημα για το διτό σύστημα εκπαίδευσης κατάρτιση στη Γερμανία που είναι ιδιαίτερο πετυχημένο αλλά επειδή ε, μειώνεται το ποστό εκείνων που επιλέγουν αυτό το σύστημα, έχουμε κάποιους προβληματισμούς πώς θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε αυτό το σύστημα. Ε, πήραμε κάποια μέτρα για να αυξήσουμε την ε, διασύνδεση μεταξύ των δύο μοντέλων. Γιατί πολλές επιχειρήσεις ε, προτείνουν ένα, ένα μοντέλο επί βάση του οποίου μπορεί κανείς να συνδυάσει την επαγγελματική κατάρτιση με ακαδημαϊκές σπουδές. Αλλά η πραγματικότητα της επιχειρήσης έδειξε ότι ακριβώς ε, ο συνδυασμός με ε, καλά καλής επαγγελματικής εξειδίκευσης με ακαδημαϊκές σπουδές είναι, μπορεί να είναι ιδιαίτερος πετυχημένη γιατί ακριβώς συνδέει τη θεωρία με την πράξη. Γι' αυτό θέλουμε να παράσουν περισσότερες δυνατότητες ε, και επαγγελματικής επιμόρφωσης. Ακόμα και αυτούς που έχουν κάνει μια επαγγελματική κατάρτιση να μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή και εντός της επιχείρησης αλλά και εξωτερικά με σπουδές στα πανεπιστήμια. Τώρα, όσον αφορά την πίζα, Στη Γερμανία για πολύ καιρό ε, θεωρεί το απορριπταίο το να συνδέεται ε, η εκπαίδευση με την ποσοτική αξιολόγηση, με την ποσοτικοποίηση, γιατί θεωρούσαμε ότι η παιδεία είναι κάτι πολύ πιο ε, σφαιρικό από τους ποσοτικούς δείκτες. Από την άλλη, ε, θα έπρεπε να αποδείξει κανείς ποια είναι τα προτερήματα των διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων. Και έτσι τα ομόσπονδα κρατήδια αποφάσισαν να υποβληθούν σε αυτή τη σύγκριση. Ε, η Υπουργό Παιδείας προτείνει εκούσια να υπάρξουν από κοινού πρωτοβουλίες, από κοινού δηλαδή μεταξύ των ομόσπονδων χωρών ε, διοργανωμένες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού επίπεδου. Αυτή είναι η προσπάθεια συντονισμού των επιμέρους εκπαιδευτικών πολιτικών. Ε, κυρία από την ε, Τσεχία μίλησε για τους ε, για τον ε, αριθμό των υπουργών. Όσον αφορά το πρόβλημα για μένα πιο σημαντική είναι η σταθερότητα της πολιτικής, η έλλειψη σταθερότητας της πολιτικής. Αυτή ορισμένες εκπαιδευτικές πολιτικές συνεχίστηκαν και με την αλλαγή της κυβέρνησης. Αλλά βεβαίως υπάρχουν προβλήματα εδώ, στο, προβλήμα, στο πλαίσιο αυτών των ε, σχολικών, των εκπαιδευτικών κλάστερς, να μπορέσουν οι μαθητές από όλες τις περιοχές να έχουν μία εκπαίδευση από τον υπηαγωγείο έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βεβαίως αυτό συνοδεύτηκε με υψηλό κόστος και ορισμένη μία υπουργός ε, παιδείας αναγκάστηκε να παραιτηθεί, αλλά εκ των υστέρων θεωρήθηκε ότι ήταν μία ε, σωστή ιδέα. Δεύτερον, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας τα τελευταία χρόνια με μικρές ε, διακυμάνσεις ε, κινήθηκε στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή τα χειρότερα χρόνια όπου η Πορτογαλία ήταν ε, υπό την αιγίδα του Δούνου του κρατήθηκε, διατηρήθηκε σταθερός παρόλα αυτά ο προϋπολογισμός, δηλαδή οι αποδοχές ε, μειώθηκαν, αλλά όχι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων. Το γεγονός ότι δεν είχαμε πολλά χρήματα, πολλά κονδύλια στη διάθεσή μας, μας υποχρέωσε να επιφέρουμε κάποιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες ε, δεν θα ήταν τα πανηρές εφόσον θέλαμε να βελτιώσουμε τα πράγματα, είμαστε υπερχομένοι να το κάνουμε χωρίς επιπρόσθετο κόστος. Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι υπήρξε ένα είδος μηχανισμού αυτορύθμισης ούτως ώστε για παράδειγμα να υπάρξουν εξωτερικές ε, αξιολογήσεις, αποτιμήσεις και τα συστήματα αυτά τα, τα τεστ αυτά, συγγνώμη, γινόντουσαν κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ε, σχολικής ε, εποχής. Και αυτό λειτουργήσε σαν κίνητρο για τους μαθητές ούτως ώστε να υπάρξει και παιδαγωγικά αλλά και μαθησιακά μια καλύτερη οργάνωση των σχολείων και αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα. Εάν δούμε τα αποτελέσματα της πίζα ε, όταν τα αποτελέσματα είναι θετικά Εάν τα αποτελέσματα είχαν εξαφανιστεί, συγγνώμη, στα σερτάρια των Υπουργών, ε, δεν θα υπήρχαν θετικές αντιδράσεις μεταρρύθμισης. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με τέσσερα ζητήματα. Καταρχάς, θα ήθελα να αναφερθώ για τις, στις εμπειρίες της Τσεχίας για την αποκέντρωση το 2000 ε, έγινε μια αρκετά μεγάλη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και δημιουργήθηκαν αυτόνομες περιφέρειες, οι οποίες ε, προ... άρχισαν ε, βεβαίως να ζητούν πολύ λογικά αρμοδιότητες σε κάποιους τομείς και τώρα το 2017 είναι τέτοια η κατάσταση που έχει 14 περιφέρειες η Τσεχία. Υπάρχουν το τοπικές και περιφερειακές αυτοδιοικήσεις. Έχουμε 14 περίπου διαφορετικά συστήματα εκπαίδευσης. Ε, γι' αυτό ε, είναι και διαφορετικές και είναι και διαφορετική η στάση των διαφορών περιφερειών. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να διατηρηθεί η ακαιρεότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. Ε, ε, βεβαίως ε, η Εθνική Επιθεώρηση της Αιγείας είναι ένας οργανισμός σε επίπεδο εθνικό που προβαίνει στην αξιολόγηση μεταξύ άλλων της ποιότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων των περιφερειών και αν είναι σωστή και η κατάρτιση των διδασκόντων. Υπάρχει ένα πρόβλημα λοιπόν με την την, ε, το συντονισμό όλων αυτών ε, των προβλημάτων που μπορεί να, να υπάρξουν ε, μεταξύ των 14 αυτόνομων περιφερειακών συστημάτων και καταλαβαίνετε και τι γίνεται κάθε φορά που υπάρχει μία αλλαγή. Υπάρχει χρηματοδότηση αναμαθητή, ανασπούδαστη. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό που του αντιστοιχεί, όμως μπορούν να διορθώσουν τα ποσά οι περιφέρειες και να επηρεάσουν τον προσανατολισμό της παιδείας ε, στην ε, εκάστοτε περιφέρεια. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα ε, πριν από το 2005 υπήρχε ένα γενικό σχήμα παιδείας ε, που ε, υπήρχε για παράδειγμα στην 6 Δημοτικού στην πρώτη Νοεμβρίου γινόταν, την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου γινόταν μια αξιολόγηση και ήταν ίδια την πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη οι μαθητές ε, ε, ε, μελετούσαν το ίδιο πράγμα σε ολόκληρη την Τσεχία. Μετά όμως... Υπήρχε ένα επίπεδο γενικό για συγκεκριμένα θέματα, για συγκεκριμένα μαθήματα τα οποία έπρεπε να διδάσκονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο ανάμεσα για παράδειγμα στη Δετάρτη και στην Έκτη Δημοτικού αλλά δεν επέβαλε σε ποια χρονική στιγμή ακριβώς έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Από τη μία λοιπόν δίνεται μια ε, ευχέρεια στα ε, σχολεία. Από την άλλη δημιουργούνται κάποιες δυσκολίες όταν ένα παιδί ε, μετακομίζει. Ένα διτό σύστημα δεν υπάρχει στην Τσεχία παρά το γεγονός ότι εμείς προσπαθούμε να υποστηρίξουμε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η άποψη των σχολείων ε, και των εργοδοτών είναι διαφορετική. Σε πολλές περιπτώσεις οι εργοδότες θα προτιμούσαν ε, τα σχολεία να τους παρέχουν ε, τους σπουδαστές που είναι σε θεωρητικό επίπεδο έτοιμοι αλλά έχουν και πρακτικές γνώσεις που θα είναι ένα τελικό προϊόν θα τους επιτρέψει να εργαστούν σε μία επιχειρήση. Υπάρχει μία μείωση ενδιαφέροντος ε, για την επαγγελματική κατάρτιση μεταξύ των σπουδαστών, ε, γιατί... Είναι πολύ, γιατί είναι πολύ χαμηλή μισθή όταν αρχίζουν να δουλεύουν ε, και προσπαθούν να προσανατολιστούν σε εντελώς διαφορετικό τρόπο από, από, από απόψεις εκπαίδευσης. Θα υπάρξει βέβαια και άλλη αλλαγή κατά τα ερχόμενα έτη λόγω των αποτελεσμάτων ε, την, ε, της ε, πίζα και βέβαια αυτό θα έχει να κάνει και με την εκπαίδευση των διδασκόντων. Υπάρχει μια συγκεκριμένη σχολή για τους διδάσκοντες ε, δεν ε, είναι επαρκή συχνά οι δεξιότητες και οι γνώσεις ενός διδάσκοντος που βγαίνει από αυτή τη σχολή διδασκόντων ώστε να μπορεί να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Οπότε θα προσπαθήσουμε να μεταρρυθμίσουμε την προετοιμασία των διδασκόντων θα δούμε ποιες είναι οι απαραίτητες δεξιότητες και των μαθητών και των σπουδαστών, αλλά και των διδασκόντων, γιατί οι διδάσκοντες δεν έχουν συχνά ε, ε, επιτυχιούχοι των, ε, των σχολών παιδαγωγικής, δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να διδάξουν τα παιδιά. Δεν γνωρίζουν την, επαρκο, την πληροφορική, για παράδειγμα, δεν γνωρίζουν ξένες γλώσσες έχουν επίσης ε, ε, λίγες γνώσεις σχέση με το πώς θα αντιμετωπίσουν ένα παιδί που έχει κάποιες μαθησιακές δυσκολίες ε, ή κάποια αναπηρία. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν και προσπαθούμε να το καλύψουμε. Θέλουμε να υποστηρίξουμε την ένταξη και θέλουμε ε, σε κάθε περίπτωση να μπορούμε να βοηθήσουμε τους διδάσκοντες να αντιμετωπίζουν ε, μία τέτοιου είδους περίπτωση ενός παιδιού με ειδικέ ανάγκες. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Όμως δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Δύο λεπτά μας μένουν. Η σημερινή ανταλλαγή απόψεων μας ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και είμαι βέβαιη ότι θα ακούσουμε πολύ περισσότερες προτάσεις όσον αφορά το σχέδιο γνωμοδότησής μας, ε, ε, το σχέδιο ε, έκθεσής μας στο πλαίσιο της ε, διευκόλυνσης εγγύησης για τους νέους, ε, την, ε, τα εκπαιδευτικά συστήματα. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις και οι ομιλίες ήταν πάρα πολύ χρήσιμες. Η εκπαίδευση αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει φτάσει η χρονική στιγμή να έχουμε πληροφορίες και μια γενική εικόνα για τα αποτελέσματα, για τις επιδόσεις των μαθητών στα σχολεία. Η έρευνα αυτή λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική, μπορούμε να αντλήσουμε πολλά συμπεράσματα, ακόμη και αν δεν υπάρχει πανάκια δυστυχώς, μπορούμε να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα γενικά, ε, όμως πρέπει για παράδειγμα να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην εκπαίδευση των διδασκόντων για να μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της αγοράς εργασίας και στις παγκόσμιες προκλήσεις. Ε, για να γίνει κάτι τέτοιο, τα κράτη-μέλη πρέπει να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές επίσης ε, πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια να αυξήσουν το κύρος και την αναγνώριση του λειτουργήματος ε, του ε, διδασκάλου. Και πρέπει επίσης και τα παιδιά να σέβονται τους διδάσκοντες. Στο πλαίσιο αυτό χρειαζόμαστε λοιπόν πολύ πολύ μεγαλύτερη συνεργασία. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που συμμετείχατε σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων και κυρίσω το πέρας της ε, πρωινής μας συνεδρίασης. Θα τα ξαναπούμε στις 3 η ώρα το απόγευμα θα πρέπει επίσης να σας ανακοινώσω ότι επειδή υπάρχει και μία ακόμη εκδήλωση ε, σε αυτή την αίθουσα, ε, μετά που θα τελειώσει η συνεδρίαση, θα ήθελα να μην, να μην αφήσετε τίποτε από τα προσωπικά σας αντικείμενα ε, στην αίθουσα αυτή, γιατί το απόγευμα θα συνεδριάσουμε σε άλλη αίθουσα.